Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Μη φοβάστε, καθίστε. Alors, nous commençons... Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας την απογευματινή μας συνεδρίαση με μία ακρόαση με θέμα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Η Επιτροπή Μεταφορών, της οποίας προεδρεύω, διοργανώνει σήμερα αυτή τη δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό και στόχος της ακρόασης είναι να τεκμηριωθεί η έκθεση πρωτοβουλίας με τον ίδιο τίτλο που θα εκπονηθεί βάσει της ανακοίνωση της Κομισιόν επί του θέματος. Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες για την έκθεση, ο εισήγητή και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών έκριναν αναγκαίο να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων με τους εμπειρογνώμονες, τους οποίους καλωσορίζω, δεδομένης της εμβέλεια ε, της ανακοίνωση και των οριζόντιων ε, και τον οριζόντιο τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τον τομέα του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν προετοιμάστηκε η ακρόαση σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και οι βουλευτές της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουν προσκληθεί να παραστούν εδώ στην ακρόαση αυτή όπως και όλοι οι ευρωβουλευτές που εργάστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τις ε, εκπομπές στον τομέα των αυτοκινήτων, η Επιτροπή που ονομάζεται ΕΜΙΣ. Η ακρόαση θα περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Περιβάλλοντος που θα μας μιλήσει για την τρέχουσα κατάσταση και θα κάνει και κάποιες προβλέψεις για το μέλλον της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών. Θα ακούσουμε και έναν ε, ερευνητή της ΕΜΦΡΑΣ που θα μας παρουσιάσει αυτό που ονομάζουμε εξωτερικά κόστη των μεταφορών, καθώς και το ρόλο των τιμών, των φόρων και των τελών επίσης. Το δεύτερο τμήμα θα εστιαστεί σε μια συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων ε, του κλάδου των κυριοτρόπων μεταφορών ε, και ο ο κύριος ομιλητής θα είναι ο κύριος Εκχάουτ, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας ε, ε, για αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας, για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Οι συζητήσει θα ακολουθήσουν το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο γύρο τραπέζης, που θα προεδρεύσει ο κύριος Εκχάουτ. Οπότε σας καλωσορίζω όλους στην Επιτροπή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι το πρώτο μέρος που είναι οι ομιλητές μας, Α, εκεί βρίσκονται. Αγαπητοί ομιλητές, έχετε 7 λεπτά ο καθένας για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας και το δεύτερο τμήμα το οποίο θα προεδρεύσει ο κ. Μπάς θα διαρκέσει λίγο περισσότερο διότι ο Μπάς Εκάουτ θα ε, προεδρεύσει ένα γύρο τραπέζι 45 λεπτών με τους εκπροσώπους του κλάδου. Καλό λοιπόν αμέσω τον κύριο. συγγνώμη, πρώτα απ' όλα. Δίνω το λόγο στον εισηγητή μα από την Επιτροπή Μεταφορών για να μας ε, παρουσιάσει το θέμα. Έχετε το λόγο κύριε Μπάσεκχαουτ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, στα εισαγωγικά μου σχόλια, διότι σήμερα είναι το πιο σημαντικό είναι να ακούσουμε τους ειδικού, τους εμπειρογνώμονε. Γι' αυτό γίνεται και η ακρόαση. Εγώ προετοιμάζω την έκθεσή μου και πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντική συζήτηση για το μέλλον των μεταφορών με χαμηλή ε, χρήση άνθρακα. Εάν δείτε στην έκθεση την περσινή του Ιουλίου, αν δείτε τον τομέα των μεταφορών, η απανθρακοποίηση είναι μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει μετά τη Συμφωνία των Παρισίων. Όλοι γνωρίζουμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε κάτω από του δύο βαθμού Κελσίου, ε, να υπάρξει μείωση δηλαδή τάξη των δύο βαθμών Κελσίου, ε, μέχρι και 1,5 και αυτό χρειάζεται προσπάθεια σε πολλού κλάδου Έχει δοθεί έμφαση σε κάποιου τομεί όπω το τομέα τη ενέργεια, όμω ε, ε, δυστυχώς και αδίκως δεν δόθηκε έμφαση στον τομέα των μεταφορών που επίσης γίνονται πολλά πράγματα. Η Κομισιόν με την ανακοίνωσή τη ε, έθεσε το θέμα αυτό στο προσκήνιο και εμεί ως Κοινοβούλιο τώρα θα πρέπει και εμείς να πάρουμε θέση. Και βεβαίως ε, αυτό που προτείνουμε τελικά θα δώσει και κατευθείας γραμμές προς την Κομισιόν ε, για να προετοιμάσει τις νομοθετικές της προτάσεις που έχει υποσχεθεί. Η πρόεδρος η κυρία Ντέλη από Καρύμα, διότι είμαι εδώ τώρα κάθομαι στη θέση αυτή και πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ε, θα έχουμε δύο παρουσιάσεις που θα μιλήσουν για όλα τα σημαντικά ζητήματα. Κάποιο από την περιβαλλοντική, Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρεσία που θα δείξει πώς ο τομέας των μεταφορών αναπτύσσεται, πώς δείχνει ότι είναι ένας από τους κλάδους όπου η απαλλαγή από τον, άνθρακο, από τον άνθρακα δεν έχει ξεκινήσει πραγματικά. Γίνονται κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει ξεκινήσει πραγματικά. Πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό στον τομέα των μεταφορών σε σχέση με τι εξελίξει με τον άνθρακα σε άλλου κλάδου. Και μετά φτάνουμε σε μια άλλη, έχουμε μια άλλη παρουσίαση, όπου έχει στο προσκήνιο ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα των τιμών. Ε, της τιμολόγησης. Είναι πάντα σημαντικό το θέμα αυτό βέβαια και σίγουρα θα αποτελέσει μέρος της συζήτησης που θα μας απασχολήσει πώς θα συμβεί αυτό ακριβώς, θα το δούμε, αλλά είναι σημαντικό αυτό και διάφορους, διάφορα μέσα μεταφοράς θα έχουμε έτσι μια σαφέστερη εικόνα. Θα ξεκινήσει λοιπόν από εκεί πέρα μια συζήτηση, ένα πάνελ για τους διάφορους Τρόπου μεταφορά τα, τα διάφορα μέσα μεταφορά, δεν μπορούμε βέβαια να έχουμε πρόσωπου από όλα τα μέσα μεταφορά, αλλά έχουμε εδώ κάποιου ε, εκπρόσωπους κλειδιά, είτε μιλάμε για οδικέ μεταφορέ, είτε μιλάμε για αερομεταφορέ, είτε μιλάμε για θαλάσσιε μεταφορέ, αλλά και βεβαίω ε, εσωτερικών υδάτων, εσωτερικών ε, θαλασσιών οδών. Εξετάζουμε λοιπόν τι γίνεται στο δικό σα κλάδο, τι έχει γίνει ως τώρα, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί και τι χρειάζεστε τι αναμένετε από τους πολιτικούς ηθήνοντες. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό ε, μία μορφή ερωταπαντήσεων ε, για να είναι έτσι κάπως πιο ζωντανή η ακρόαση. Ιδάλλως ε, έχουμε μόνο έτσι, μακροσκελείς μονολόγους. Θα σταματήσω λοιπόν το, το δικό μου μονόλογο διότι αυτό που έχει ενδιαφέρον όπως είπα και στην αρχή είναι αυτό που θα πούνε οι εμπειρογνώμενες, όχι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί πάντα δυσκολεύονται να μην πάρουν το λόγο, αλλά σήμερα ε, πρωταγωνιστούν και μας κατευθύνουν οι εμπειρογνώμονες. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ δεν θα τον πω με το μικρό του, θα τον πω με το επίθετο. Ξεκινάει λοιπόν αυτός ο πρώτος, η πρώτη στρογγυλή τράπεζα με τους εμπειρογνώμονες ως πρώτα ο κύριος Αλφρέντο Σάνσεθ Βιθέντε, είστε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και έχετε 7 λεπτά για την παρουσίασή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πρόσκληση που μου απίφθινε και τη διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης και που μας κάλεσε να σας δώσουμε κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τις μεταφορές και το περιβάλλον. Είναι χαρά μου λοιπόν που βρίσκομαι εδώ. Έχω φέρει μαζί μου και μια παρουσίαση με διαφάνειες για να μας ε, οδηγήσει. Αλφρέδο Σάντζες Φιθέντε, ονομάζομαι, εργάζομαι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στην ε, Κοπενχάγη. Θα ήθελα να επισημάνω πόσο κρίσιμη σημασία είναι να γίνει κατανοητή η σημασία των εκπομπών των μεταφορών στο περιβάλλον και στην υγεία. Πρόκειται για ένα περίπλοκο σύστημα ε, διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων ε, ανάμεσα στις εκπομπές, ε, τις τα ρηπογόνα αέρια, αλλά και τις επιπτώσεις των εκπομπών αυτών στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και στο, στα οικοσυστήματα και στο κλίμα. Για την ανθρώπινη υγεία η μόλυνση, η ρήπανση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ε, ε, για την ε, θέση της υγείας του ανθρώπου σε κίνδυνο και την μείωση του προσδόκιμου ζωής. Και η αυξήσεις, η αύξηση των, ε, της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα επίσης αποτελούν έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης ανθρώπινης υγείας. Επίσης περιβαλλοντικά έχουν επιπτώσεις με πλημμύρες, βροχοπτώσεις, ε, αυξημένες βροχοπτώσεις κτλ. Έτσι λοιπόν ε, οι εκπομπές επηρεάζουν αρνητικά τόσο το περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη υγεία. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε λοιπόν ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές δεν είναι μόνο εκπομπές αλλά και ο θόρυβος για παράδειγμα. Μιλώντας για την ποιότητα του αέρα, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πολιτικές για την ποιότητα του ε, αέρα έχουν αποφέρει αποτελέσματα, έχουν βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις πόλεις μας, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Όπως βλέπετε εδώ στο χάρτη, όπου μιλούμε για το διοξίδιο του αζότου, το οποίο είναι ε, ένας ε, ρηπογόνος παράγοντας, ε, αέριος ρηπογόνος παράγοντας που συνδέεται άμεσα με τις, με τις εκπομπές. Οι κόκκινες βουλίτσες που βλέπετε είναι τα γεωγραφικά σημεία όπου τα όρια αυτής της ουσίας βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από τα επιτρεπτά. Γύρω στα 60% ε, του διοξιδίου του αζότου προέρχεται από τις οδικές μεταφορές και σε κάποιες χώρες είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό, 80% ή και παραπάνω. Οι υψηλέ εκπομπές λοιπόν ε, διοξιδίου του αζότου επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα, του αέρα και ε, οφείλονται, σε αυτές οφείλονται και το γεγονός ότι πολλές χώρες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν τεθεί από τους ε, ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ποιότητα του αέρα. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ε, ότι ε, έχει αρχίσει μια διαδικασία εφαρμογής πολιτικών για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι μεταφορές λοιπόν ε, ευθύνονται για το 1 τέταρτο όλων των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ε, διότι βλέπετε και εδώ στο γράφημα ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 1990. 20% έχουν, έχουν αυξηθεί τα, η τάση αυτή άρχισε να αντιστρέφεται το 2007 όταν άρχισαν να γίνονται αισθητέ και οι επιπτώσεις ε, της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, το 2014 και το 2015, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε συλλήξει, οι ε, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πήραν και πάλι την ανιούσα. Οι προβλέψεις για τις εκπομπές αερίων, σύμφωνα με τα κράτη-μέλη, σύμφωνα και με τις εθνικές πολιτικές που έχουν ε, ήδη τεθεί σε εφαρμογή, δεν φαίνεται ότι θα μειώσουν ε, το πρόβλημα σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έχουν δεσμευτεί στον στόχο ε, μείωσης ε, των ε, εκπομπών που προέρχονται από τις μεταφορές κατά 60% έως το 2050. Βλέπετε εδώ στο γράφημα πόσο μεγάλο, μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση. Χρειάζεται δηλαδή να μειώσουμε κατά 67% τις εκπομπές προκειμένου να επιτύχουμε απλώς αυτό το στόχο. Οι οδικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθούν ε, τα επόμενα χρόνια κατά 40% έως το 2050. Γι' αυτό το λόγο η βασικότερη πρόκληση είναι να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις και να τις συνδυάσουμε με όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για μεταφορές. Όπως και στο παρελθόν, ε, οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, τελικά υπερσκελίζονται από το γεγονός ότι αυξάνεται δυσανάλογα πολύ η ζήτηση για μεταφορές. Η ενέργεια που χρειάζεται να δαπανίσει κανείς για την ε, διάνυση 100 χιλιόμετρων έχει μειωθεί γιατί τα, τα οχήματα είναι πλέον πιο αποδοτικά Ωστόσο, έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός των, ε, των οχημάτων που κυκλοφορούν και έτσι αυξήθηκαν τα επίπεδα διοξιδίου του, του άνθρακα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καλές προοπτικές τα ε, αυτοκίνητα να απαλλαγούν σύν το χρόνο από την ε, κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, αυτό δεν ισχύει για όλους τους τρόπους ε, μεταφορών. Γι' αυτό απαιτείται ένας ριζοσπαστικός τρόπος αλλαγής ε, ε, του τρόπου με τον οποίο μετακινούμαστε. Ε, να σας δώσω τώρα κάποια στοιχεία. Οι μεταφορές ευθύνονται για το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταφορές είναι ο μοναδικός κλάδος της οικονομίας που ευθύνεται για μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ε, ε, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν σημειώσει πρόοδο, χωρίς όμως να μπορούν να αντισταθμίσουν την αυξημένη ζήτηση και χρειάζονται πιο ριζοσπαστικές λύσεις αν θέλουμε ε, τα επόμενα χρόνια να επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σάντσες. Τηρήσατε το χρόνο σας, κάντε το ίδιο παρακαλούμε και εσείς κύριε Ντανιλ Σότερ, το λόγο. Okay, Καλημέρα. Daniel Σούτερ από το Ινστιτούτο Ίνφρα στην Ζηρίχη ε, όπου ε, εργάζομαι στο τμήμα εξωτερικών, ε, εξωτερικού κόστους των μεταφορών και έπειτα από αυτήν την εποπτεία που μας δόθηκε θα ήθελα εγώ να σας παρουσιάσω τα εξωτερικά κόστη των μεταφορών. Τι είναι αυτά. Πρόκειται για ε, κόστη τα οποία προκαλούν οι συμμετέχοντες ε, στις μεταφορές αλλά δεν αναλαμβάνονται από εκείνους που ε, πραγματοποιούν τις μεταφορές. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε λόγο για αποτυχία της αγοράς. Πολύ συχνά συνδυάζεται το φαινόμενο του κόστους των μεταφορών με ε, την ε, διεθνοποίηση ε, η οποία ωστόσο μπορεί και να αποτελέσει μια δυνατότητα για μείωση του κόστους. Ποιες, ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που μας ενδιαφέρουν. Πρόκειται για ε, κόστος υγείας, απώλειες παραγωγικότητας, βλαβών και ζημιών στα οικοσυστήματα, ή ε, βλάβες και ζημίες σε κτήματα ή και άειλες ζημίες. Πέντε είναι οι βασικότεροι τομείς. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφορούν κυρίως ε, την ε, ρήπανση του αέρα, η κλιματική αλλαγή και ο θόρυβος. Επίσης υπάρχουν σημαντικά, σημαντικά κόστη που προκύπτουν από τα ατυχήματα. Αυτό λοιπόν είναι το συνολικό εξωτερικό κόστος των μεταφορών στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι ε, το κόστος αυτό ανέρχεται σε περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια ε, ευρώ και ευθύνονται για το κόστος αυτό κατά 90% και πλέον οι οδικές μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε δεδομένα του 2008 υπάρχει, ε, υποθέτουμε ότι έχουν αλλάξει ε, ε, έκτοτε τα πράγματα, ε, έχει βελτιωθεί η τεχνολογία, ωστόσο αυτή ενδέχεται να έχει αντισταθμιστεί από την αύξηση της ζήτησης. Ε, όπως βλέπετε εδώ στο γράφημα, βλέπετε τις, ε, το, το κόστος για τις εμπορευματικές μεταφορές, αριστερά βλέπετε τις, ε, ε, τα φορτηγά, τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και στο, στα δεξιά τις εσωτερικές πλούτες οδού. Το κόστος της, των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αν είναι τέσσερα, τέσσερις φορές μεγαλύτερες, ε, μεγαλύτερο από τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αν και υπάρχει μια εσωτερική διαβάθμιση και διαφοροποίηση στις σιδηροδρομικές μεταφορές, είναι άλλο το κόστος των ηλεκτρικών σιδηροδρομικών μεταφορών και άλλο των ε, πετρελαιοκίνητων σιδηροδρομικών μεταφορών. η, εσωτερικοποίηση του κόστους ε, του εξωτερικού κόστου στην Ευρώπη έχει ήδη επιχειρηθεί να υλοποιηθεί, ωστόσο όχι με επαρκή τρόπο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει ε, εδώ και λίγο καιρό ε, στα διόδια ένα μέρος των διοδίων που ε, χρησιμοποιείται και που επιβάλλεται ως τέλος για την αντιστάθμιση των αρνητικών περιβαλλοντικών υποπτώσεων στην ποιότητα του αέρα. Ταυτόχρονα μέσω των διοδίων μπορεί να, μπορεί να καλυφθεί και ένα μέρος του κόστους που σχετίζεται με τα ατυχήματα. Αντίστοιχες, ε, αντίστοιχα τέλη ε, επιβάλλονται και στις ε, αεροπορικές μεταφορές και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Οι επιπτώσεις της εσωτερικοποίησης του εξωτερικού κόστους μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών. Επίσης, μια τέτοια εσωτερικοποίηση μπορεί να οδηγήσει και σε εξυγίαση των δημοσιονομικών μιας χώρας. Και ε, ε τελευταίο, ε, μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση ε, της ζήτησης για οδικές μεταφορές. Τα διόδια στην Ελβετία δείχνουν ότι οδήγησαν σε σχεδόν 25% μείωση των οδικών μεταφορών και αντιστοίχω μειώθηκαν και οι εκπομπέ. Βεβαίω αυτό το παράδειγμα δείχνει επίση ότι η εσωτερικοποίηση εξωτερικού κόστου δεν αρκεί πάντοτε για, την επίτευξη πολιτικών στόχων, πολιτικών περιβαλλοντικών στόχων. Εδώ σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της ε, Ελβετίας υπάρχει ένα άρθρο για την προστασία ε, των Άλπαιων που ε, ε, ορίζει ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία 65.000 οχημάτων κατ' στην Ελβετία. Δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πάντως ε, διαγράφεται εδώ και χρόνια μια θετική τάση. Να σας πω και δύο λόγια για τις προκλήσεις. Στην βάση της, της, ε, των επιστημονικών ε, δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, η DG Move θα εκπονήσει σύντομα μια μελέτη σχέση με την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους και θα αφορά όλες τις χώρες και όλους τους τρόπους μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική για την κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές ε, είναι ένα σημαντικό θέμα που θα τροφοδοτηθεί ε, και από αυτήν την μελέτη. Ε, ιδίως ε, όσον αφορά διαστάσεις που αφορούν το κλίμα και τα ατυχήματα. Επίσης, χαιρετίζουμε από τη δική μας πλευρά την χάραξη μιας τέτοιας στρατηγικής. Ωστόσο, απαιτούνται και άλλα ρυθμιστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα ο ορισμός ανώτατων ορίων εκπομπών. Και γι' αυτό προσβλέπουμε και στα λεπτομερή στοιχεία που, στα οποία θα καταλήξει ε, η στρατηγική αυτή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σούτερ. Για να μην χάνουμε λόγο χρόνο, δίνω τον λόγο στο συντονιστή μας κύριο Μπάς Έικχαουτ για το δεύτερο τμήμα του γύρου τραπέζης. Κύριε Μπάς Έικαουτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο πάνελ συζήτησης και μετά θα ακολουθήσουν 45-50 λεπτά για ερωταπαντήσεις. Μετά από αυτό το γύρο δηλαδή. Έχουμε έξι εμπειρογνώμονες, έξι εκπροσώπους διαφόρων ε, τρόπων ε, μεταφορών, για να το πω έτσι. Θα μας πούν τι συμβαίνει στον τομέα τους. Λοιπόν, να σας τους παρουσιάσω. Πρώτα απ' όλα στα δεξιά έχουμε τον Ερικ Ζωνάρ, Γενικό Γραμματέα ε, της γνωστής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Στα αριστερά του έχουμε τον Ματίας Μέιτζ, Μέιτζε, συγγνώμη, ήταν το πιο δύσκολο όνομα για να το προφέρω, Γενικό Εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών. Μετά έχουμε από τους ελβετικούς σιδηροδρόμους έναν εμπειρογνώμονα, τον Μίχαλ Μπέσ. Και μετά από την Airbus, για να περάσουμε στην αεροπορία, ε, έχουμε δηλαδή τις οδικές μεταφορέ σιδηροδρομικές και μετά την αεροπορία ε, και από την Airbus έχουμε τον Τιερή Νόβατσικ, ε, Διευθυντή Ευρωπαϊκών ε, Θεμάτων και μετά περνάμε στα νερά, στα ύδατα και έχουμε δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Κάριν Τεσχέπερ, Διευθύντρια του Inland Navigation Europe, ε, αφορά φυσικά την εσωτερική ναυσιπλοεία και μετά έχουμε τον Πάτρικ Φερχούβεν, Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλοίοκτητών για να πάμε στους ωκεανούς, για να το πω έτσι. Αυτή είναι η διάφοροι εμπειρογνώμονες που έχουμε και ξεκινάμε με τον κύριο Ζωνάρ, Ε, λοιπόν, έχοντα ακούσει τώρα τι διάφορε ιστορίε που ακούσαμε και τον Ντάνιελ Σάτερ που μίλησε για τα εξωτερικά κόστη, που φαίνεται να είναι υψηλότερα για τι οδικέ μεταφορέ αυτή τη στιγμή, ίσω είναι καλύτερο ξεκινώντα να μα πείτε ποιε είναι οι εξελίξει που βλέπετε εσεί, ειδικότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η κατασκευή αυτοκινήτων βάσει του παρελθόντο και των πιο πρόσφατων εξελίξεων, πώ βλέπετε τι προοπτικέ. Ευχαριστώ. Πώς βλέπουμε εμείς το μέλλον στην αυτοκινητομηχανία για να συνεισφέρουμε ε, σε μια κινητικότητα με χαμηλή χρυσή άνθρακα. Πέντε είναι οι πυλώνες. Πρώτον, και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, εμείς επικεντρωνόμαστε έτσι ώστε τα τεστ για τις εκπομπές να γίνονται με το σωστό τρόπο. Δηλαδή πάμε στην WRTP για το πώς θα μετράμε τις εκπομπές, το συντομότερο δυνατόν. Το Σεπτέμβριο του 2017 ήδη φέτος για τα νέα οχήματα, ε, όμως από το Σεπτέμβριο του 2018. Αυτό είναι το πρώτο. Οι δοκιμές λέει τα τεστ. Δεύτερον, το θέμα των καυσίμων ε, και της καύσης ε, μέσω ε, των, κινητήρων καύσης, εν περιπτώσει. Υπάρχουν πολλές κριτικές. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι θα εξαλίσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να γίνει όσο γίνεται καλύτερη η, η χρήση αυτού του συστήματος και θέλουμε επίσης να, να χρησιμοποιούμε τον ντίζελ αλλά με έναν τρόπο που να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Τώρα, εναλλακτικά συστήματα μετάδοσης κίνησης για να οδηγηθούμε σιγά σιγά σε μηδενικές εκπομπές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τι δυνατότητε που έχουμε σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών και τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί πέρα σε επίπεδο βιοκαυσίμων. Ξέρω ότι δεν είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Θα πρέπει όμω να δούμε και τα βιοκαύσιμα δεύτερη γενιά και θα πρέπει να υπάρξει μια σαφήνεια από του πολιτικού θύνοντε. Φυσικό αέριο. Μια άλλη δυνατότητα για τη μείωση των εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα. Και από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τι μηδενικέ εκπομπέ, εξετάζουμε ποιε, ποιες είναι οι δυνατότητες που μας, προσφέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα. Το τέταρτο τώρα. Πρέπει να υπάρξει μια μόχλευση στις δυνατότητες που μας προσφέρει η ψηφιοποίηση για πιο αποτελεσματικές ε, λύσεις. Ε, η τεχνολογία διασύνδεσης ε, μας δίνει νέες δυνατότητες όλα αυτά. Το λέει και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ένα άμεσο ε, πρώτο βήμα για να κινηθούμε σιγά σιγά ε, προς την ε, αυτόνομη οδήγηση. Και το πέμπτο που ήθελα να φέρω είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η κινητικότητα ως υπηρεσία. Το να μοιραζόμαστε αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη, το car sharing. Πρόκειται βεβαίω για κάτι καινούριο, ε, παθαίνω έδαφος, αλλά πολλοί αρχίζουν να εξετάζουν ποιες είναι οι δυνατότητες που μας παρέχει αυτό το νέο επιχειρησιακό μοντέλο πάντα στα πλαίσια του στόχου της ε, λιγότερης ε, χρήσης άνθρακα. Να δώσω μια συνέχεια σε αυτό που είπατε. Το τρίτο στο οποίο αναφερθήκατε για τις εναλλακτικέ όταν μιλήσατε για οχήματα ε, χαμηλών εκπομπών και πώς θα περάσουμε σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, ε, δεν υπάρχει ένας κίνδυνος αυτή η μετάβαση να οδηγήσει ε, στο ε, να εγκλωβιστούμε στα οχήματα μικρής ε, κατανάλωσης μικρών εκπομπών και να μην πάμε ποτέ στην, στις μηδενικές εκπομπές. Ναι, ακούστε, χρειαζόμαστε μια μεταβατική φάση. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τη σημερινή κατάσταση στο 100% σε μηδενικές εκπομπές. Θα χρειαστεί μια μεταβατική φάση. Γι' αυτό και εμείς στον κλάδο εξακολουθούμε να ζητούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε δίζελ το οποίο όμως να συμμορφώνεται με τους κανόνες, με τις προδιαγραφές. Διότι όταν μιλάμε για αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών και διότι όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά οχήματα, για ηλεκτρονική ε, με μεταφορές, θα αλλάξει τελείω το μοντέλο το επιχειρησιακό. Χρειάζεται, ε, θα πρέπει να γίνει μια ε, πολύ σημαντική αλλαγή στον τρόπο παραγωγής, θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, αυτό θα, θα επηρεάσει και τις θέσεις απασχόλησης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ε, με μιας επαναστατικά. Θα πρέπει να γίνει σταδιακά. Και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που χρειάζονται, υπάρχουν κάποιες χώρες που θέτουν κάποιους στόχους σε ό,τι αφορά τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές που εξετάζονται από την κάθε χώρα. Ε, τι είδου πολιτικές θεωρείτε εσείς ε, η οργάνωσή σας ε, είναι πιο σοφές, αν θέλετε, για να λάβει η χώρα αυτή η μετάβαση. Ακούστε, πρώτα απ' όλα, εμείς είμαστε υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, σφαιρικής. Θα πρέπει να το δούμε όχι μόνο από την άποψη των οδικών μεταφορών, πρέπει να το δούμε γενικότερα για όλου του τρόπου, για όλα τα μέσα μεταφορά. Χρειαζόμαστε επίση μια συνεπή πολιτική σε ό,τι αφορά την ε, κλιματική αλλαγή και την ποιότητα του αέρα διότι επικεντρωθήκαμε πολύ στην κλιματική αλλαγή χωρίς να μιλήσουμε αρκετά για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Θα πρέπει να το δούμε αυτό λοιπόν ολοκληρωμένα, συνολικά. Και επίσης χρειάζεται περισσότερο συντονισμός ε, και εντός της κάθε χώρας και μεταξύ των χωρών. Σε ό,τι φορά το ο καθένας, Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικέ πρωτοβουλίε κάθε, που παίρνει κάθε πόλη και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε άλλα, άλλου τύπου οχήματα ανάλογα με την πόλη. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή. Επίσης, τεχνολογική ουδετερότητα, διότι εάν θέλουμε τελικά να έχουμε ε, συστήματα κινητικότητας, συστήματα μετακίνησης, μεταφορών με μηδενική χρήση άνθρακα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Ε, Υπάρχουν πολλέ και διάφορε δυνατότητε. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα λοιπόν στου μηχανικού μας να βρουν την καλύτερη. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι η μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα. Θα γίνουν πολύ σημαντικέ αλλαγέ. Πρέπει να μπορέσουμε να τι προγραμματίσουμε. Ιδιαίτερα όταν οι στόχοι μα είναι φιλόδοξοι. Το τέταρτο σημείο είναι η ανανέωση του στόλου. Εάν δείτε σήμερα αυτή τη στιγμή τι εκπομπέ, 5% του στόλου είναι νέα οχήματα με τις νέες τεχνολογίες. Τα 95% είναι παλιά οχήματα, χωρίς αυτή, αυτή την τεχνολογία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να προωθήσουμε την ανανέωση του στόλου για να μπορέσουν να ε, έρθουν αυτές οι νέες τεχνολογικές ε, λύσεις στην αγορά. Επίσης θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στις υποδομές ε, ε φόρτωσης των ε, οχημάτων. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές, δεν θα, υπάρξει, δεν θα υπάρξει η εμπιστοσύνη για, του καταναλωτή για να κινηθούν προς τέτοιου οχήματα. Και όχι μόνο ε, ε, σε δημόσιους χώρους, στις, ε, στους αυτοκινητόδρομους, στις εθνικές οδούς, πρέπει να δούμε πώς θα επενδύσουμε και σε εμπορικά κτίρια, αλλά και πλέον στα, στις κατοικίες στις ιδιωτικές. Επίσης, οι δημόσιες προμήθειες μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να ενθαρρύνουμε την μετακίνηση προς καθαρότερα οχήματα. Έβδομο, είναι και έχω πολλά ακόμα. Ε, χρειάζεται ένα πολιτικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο πολιτικής μάλλον, το οποίο να είναι σαφές, να είναι σαφέστερο προς περιπτώσει για την ε, αφαίρεση του άνθρακα. Παραδείγματος χάρη τα βιοκαύσιμα. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα όριο για την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων, δεν μιλάμε πια για αυτά, αλλά έχουμε τη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες και θα τα χρειαστούμε αυτά ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα φορτηγά ε, και τα ε, οχήματα βαρέων κυβικών. Λοιπόν, επειδή είστε εμπειρογνώμονας για τα εναλλακτικά καύσιμα, ε, σε ό,τι φορά τη μετάβαση στις οδικές μεταφορές, ε, πόσο γρήγορα, διότι βεβαίως ε, όλοι καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, αλλά ακούσαμε ότι θα πρέπει να πάει στο μείον 60% ε, έως το 2050. Έτσι, ο τομέας των δικών μεταφορών. Πώς βλέπετε να ε, συνδυάζονται αυτά τα δύο στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Εκχάουτ, κύριε Ντελή, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω εκ μέρους ε, του Διεθνου, της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών. Άκουσα πολλά θέματα για τα οποία για να απαντήσει κανείς δεν ήθελε πολύ χρόνο, αλλά καταλαβαίνω την προσέγγιση και θεωρώ ότι είναι χρήσιμη. Ας δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε ενδεχομένω, διότι η IRU και τα μέλη μας από ολόκληρο τον κόσμο εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες οδικών μεταφορών, εκατοντάδες εκατομμύρια καθημερινών διαδρομών και πελατών ε, και έχουμε κοινωνική ευθύνη και ανησυχώ όταν ακούω ότι οι εκπομπές εξακολουθούν να αυξάνονται ε, ενώ ουσιαστικά στο δικό μας τομέα μειώνονται γιατί εγώ εκπροσωπώ τις εμπορικέ ε, δραστηριότητες τα ταξί, τα πούλμαν, τα λεωφορεία, τα φορτηγά και υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ των επιβατικών αυτοκινήτων και των εμπορικών οχημάτων. Και αυτό συχνά δεν ακούμε στις πολιτικές συζητήσεις η αγορά για τις οδικές μεταφορές. Είναι πολύ διαφοροποιημένη και πολυμορφική. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε για να δούμε πώ θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τι εμπορικέ υπηρεσίε που ήδη προσφέρει ο κλάδο μα σήμερα. Αναφέρθηκα στην κοινωνική ευθύνη του κλάδου μα. Αλλά πρώτα απ' όλα οι δραστηριότητες μας είναι επικερδείς και οι φορείς καθημερινά ε, οι επιχειρήσεις σκέφτονται πώς θα κερδίσουν χρήματα με τον πλέον περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο αλλά και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Εκτιμάμε την πρόσκληση αυτή για ε, να συζητήσουμε την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και ε, θέλω να αναρωτηθούμε, υπάρχει κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Ε, δεν θα έπρεπε να μιλήσουμε για τις εκπομπές ε, κύκλου ζωής, ε, ε, για το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Αυτό θα ήθελα να συζητήσουν οι εταιρείε και δεν συζητείται επαρκώς. Λοιπόν, ε, ξέρετε, ο κλάδος μας είναι περισσότερο από το Dieselgate και από τα γιοταχή. Ε, για παράδειγμα, το τομέας των Πούλμαν. Αν θέλετε να μετακινήσετε 50 ανθρώπου με ένα Πούλμαν, ε, καταναλώνετε κάτω από 30 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Αν πάρετε επιβατικά αυτοκίνητα, είναι τριπλάσιος, τριπλάσια η κατανάλωση, 90 με 100 λίτρα οι εταιρείε μα ενδιαφέρονται να μειώσουν την ε, κατανάλωση καυσίμων για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα, για να κάνουν οικονομία. Ε, οπότε μας ενδιαφέρει να περάσουμε σε χαμηλότερες εκπομπές και σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ε, στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Αν αναρωτιέστε τι έχει γίνει στον κλάδο μας, πρέπει να σκεφτείτε ότι επενδύουμε σε οχήματα που οι ε, εταιρείε μας πρέπει να διατηρούν για αρκετά χρόνια στο στόλο τους 6, 8, ε, και όταν μιλάμε για την κατάσταση του στόλου, θυμηθείτε ότι εμείς στον τομέα των φορτηγών, για παράδειγμα, ε, λειτουργούμε ήδη 30 με 40% οχήματα Euro 6 ήδη σήμερα και το ποσοστό αυτό είναι 20% στα Pullman. Ε, και ξέρετε τι, είναι, αν με ρωτήσετε είναι εφικτό να έχουμε 100% Euro 6 οχήματα μέχρι το 2020 θα έλεγα ναι, αλλά είναι λίγο φιλόδοξο. Οπότε όταν μιλάμε ε, πώς θα σκεφτούμε πέραν του ντίζελ, ο δικός μας κλάδος είναι υπέρ της εξέλιξης αυτής και θα την υποστηρίξουμε. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι η εγκατάλειψη του ντίζελ και αν αφήσουμε τον ντίζελ και μιλήσουμε για αναλλακτικά μεταβατικά καύσιμα και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι επίσης κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε όλες τις εναλλακτικέ που θα μείνουν ή θα ε, ε, εξαφανιστούν από την αγορά ε, πρέπει να το συζητήσουμε. Ξέρετε, είναι δύσκολο να πείσει κανεί τι εταιρείε να αγοράσει μια τελείω διαφορετική τεχνολογία χωρί να ξέρουν αν θα πιάσει τελικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει κανεί να χρησιμοποιεί ανανεώσιμε ε, μορφέ ενέργεια ή την ηλεκτροκίνηση. Ε, δεν υπάρχει μόνο η μπαταρία, τα ηλεκτρικά, ε, μπορεί να μετατρέψει κάνει τον ηλεκτρισμό σε συνθετικό μεθάνιο, υπάρχουν ε, εναλλακτικά καύσιμα, υπάρχουν πολλά πράγματα. Ας μην κοιτάμε μόνο ε, τις εξατμίσεις, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ξέρετε, μηδενικέ εκπομπές δεν σημαίνει αυτό που νομίζουμε, αλλά όλα έχουν μια τιμή, ε, το, την οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι, οι επιχειρήσεις. Ε, άκουσα για του εξωτερικού παράγοντε, πιστεύω ότι ο δικός κλάδος ήδη χρεώνεται τα περισσότερα. Είμαι, θα με ενδιαφέρον να δω τι επόμενε μελέτε που θα εμφανιστούν για να καταλήξουμε στα νούμερα όσον αφορά τι οδικέ μεταφορέ. Έχουμε ήδη υποστεί το μεγαλύτερο φόρτο και είμαι περίεργο να ακούσω από του άλλου κλάδου ε, να μου πούν πώ μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Χρειαζόμαστε τι οδικέ μεταφορέ. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο. Ε, ε, χρειαζόμαστε βασικά όλε τι τρόπου μεταφορά, αλλά με, καλύτερη, με καλύτερο τρόπο χρήση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. επίκειται μια συζήτηση για, τα, για τις προδιαγραφές όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα για τα φορτηγά. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν και ιδιαίτερα καινοτόμα ή πρωτοπόρα στον τομέα αυτών. Ε, στις ε, ΗΠΑ, ωστόσο, έχει ήδη καταρτιστεί μια τέτοια ε, πολιτική. Εσείς τι πιστεύετε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι στην πρωτοπορία στις οδικές, στις οδικές μεταφορές. Νομίζω ότι έχουμε ε, ηγετικές ικανότητες και στις οδικές μεταφορές και όσον αφορά την ε, ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης νομίζω ότι εδώ δεν βρίσκονται στην κορυφή η ΙΠΑ αλλά η Κίνα. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε μια εφικτή λύση Πράγματι, και ο υπόλοιπο κόσμο προχωρά στη μείωση των εκπομπών. Αλλά νομίζω ότι η Ευρώπη ε, έχει ε, ε, θέσει στον εαυτό τη υπερβολικά φιλόδοξου στόχου. Θέλουμε να κινηθούμε προ την ίδια κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο εφικτό. Μα ανησυχεί και μα ενδιαφέρει ταυτόχρονα η συζήτηση για τι προδιαγραφέ για το διοξίδιο του άνθρακα. Ωστόσο, πρέπει να σα πω ότι ε, στην περίπτωση των, ε, πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Στα ταξί, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι πράγματι είναι ε, πολύ χρήσιμη η εφαρμογή τέτοιων προδιαγραφών. Δεν ισχύει απαραίτητο το ίδιο και για τα επιβατικά οχήματα. Οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν, αλλά με έναν τρόπο που θα διατηρήσει και θα διαφυλάξει τον κλάδο χωρίς να, τους, ε, να, να εξοντώσει οικονομικά τις επιχειρήσεις μας. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να ε, επιδιώκουμε ε, εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν στην πράξη. Γι' αυτό και είμαστε στη διάθεση όλων των υπόλοιπων εμπλοκόμενων φορέων για συνεργασία, για συζήτηση. Πρέπει βεβαίως να καταρτιστούν προδιαγραφέ για το διεξίδιο του άνθρακα, αλλά χρειάζεται να βασιστούμε στη συζήτηση αυτή σε πραγματικά στοιχεία και να, γίνει, να χαραχτούν πολιτικές οι οποίες θα είναι εφικτές. Ευχαριστώ. Να δώσω ε, τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο των σιδηροδρόμων, τον ε, κύριο Μπες από την Ελβετία. Πώς βλέπετε εσείς την ε, τροπική μεταστροφή ε, την αλλαγή όσον αφορά τις, ε, τους τρόπους μεταφορών. Ε, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θα ε, επικεντρωθώ και θα σας δώσω την, την οπτική των σιδηροδρόμων. Νομίζω ότι οι διατροπικές μεταφορές είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει πραγματικά να τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής μας. Χρειάζονται μέτρα για να επιτύχουμε ε, τις διατροπικές μεταφορές. Ο προηγούμενος ε, ομιλητής ε, παρουσίασε ήδη το μοντέλο της ε, Ελβετίας όπου υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι ε, όσον αφορά την μείωση των ε, βαρέων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους. Έχουμε επιτύχει ορισμένα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο δεν επαρκούν, χρειάζονται ακόμη περισσότερα. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι χρειάζεται η προσαρμογή της υποδομής που έχει η κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στην, Ελβετία ε, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το διαλπικό, ε, το οποίο ε, επιτρέπει την μεταφορά, τη μετάβαση μάλλον από, την, τον έναν τρόπο μεταφοράς σε κάποιον άλλον. Άλλο θέμα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να φορτίσουμε τίζουν τα αυτοκίνητά τους οι οδηγοί ε, καθοδόν και στη συνέχεια να μπορούν ενδεχομένω να επιβάζονται σε σιδηροδρόμους για τη συνέχιση της ε, διαδρομής τους ε, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις να επιλέγουν σε κάθε περίπτωση τον βέλτιστο τρόπο μεταφοράς ε, ανθρώπων και εμπορευμάτων. because you Μιλήσατε για επενδύσεις ε, στις υποδομές που σχετίζονται και με την ε, συνδεσιμότητα. Ωστόσο υπήρξε και μια συζήτηση για το εξωτερικό κόστος και την εσωτερικοποίησή του. Εκεί υπάρχει κάποιος ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει η, ε, η πολιτική. Ναι, είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Να ενταχθεί δηλαδή ε, το εξωτερικό κόστος, αυτό που εξωτερικεύεται τόσα χρόνια στην, στον ίδιο τον τρόπο μεταφοράς. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, λέει ο Προεδρεύων, γιατί ε, είναι πάντοτε ένα πολύ αμφιλεγόμενο και ακαθόδε ζήτημα από ευρωπαϊκής προοπτικής. Αυτή η ε, εσωτερικοποίηση του κόστους, πώς ε, την ε, αντιμετωπίζετε εσείς και πώς προσέρχεστε εσείς σε αυτήν την ε, συζήτηση. Απευθύνομαι στον εκπρόσωπο των οδικών μεταφορών κυρίως. Ναι, είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους τρόπους μεταφορών. Αναφέρθηκε και, και νωρίτερα και να υπενθυμίσω ξανά ότι όταν ε, ε, εφόσον μάλλον οι οδικές μεταφορές ήδη πληρώνουν το εξωτερικό κόστος το οποίο προκαλούν, τότε θα πρέπει αυτό να ισχύσει και για τους άλλους τρόπους μεταφορών. Μας εκπλήσει, ήδη χρεωνόμαστε ε, ήδη τεράστια ποσά για την αντιστάθμιση του εξωτερικού κόστους ε, αυτού, εγώ θα έλεγα ε, ή όλοι ή κανείς. Ε, αν δείτε για τον τρόπο με τον οποίο, τον τρόπο με τον οποίο ε, είναι οργανωμένες οι οδικές μεταφορές σήμερα και το πόσο χρεώνονται ε, μέσω φορολογία, για παράδειγμα ή άλλων τελών ε, υπάρχει, υπάρχουν τα τέλη ταξινόμησης, υπάρχουν τα τέλη κυκλοφορίας ε, το ερώτημα είναι τι συμβαίνει με όλους αυτούς τους φόρους. Πράγματι χρησιμοποιούνται όλοι αυτοί οι φόροι ε, για να γίνουν επενδύσεις ε, στο δικό δίκτυο ή γίνονται επενδύσεις για να βελτιστοποιηθούν οι τρόποι μεταφοράς. Όταν λοιπόν γίνεται λόγος για ακόμα περισσότερους ε, φόρους, μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ε, θα αξιοποιηθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η εφορολογία εξακολουθεί να είναι εθνική αρμοδιότητα, Οπότε ε, βλέπουμε διάφορες πρωτοβουλίες να αναδύονται από εδώ και από εκεί. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει μια πιο ενιαία κατεύθυνση και από αυτή την άποψη θέλω να ξανατονίσω στην ανάγκη ύπαρξης κινήτρων στην Ευρώπη ώστε οι πολίτες να αγοράσουν πιο καθαρά οχήματα. Υπάρχουν διάφορα καθεστώτα και συστήματα και μηχανισμοί που συντείνουν προς αυτό ή που διευκολύνουν μια τέτοια διαδικασία. Αλλά έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα. Αν λοιπόν υπάρξει ένα πανευρωπαϊκό κίνητρο ώστε να καθοδηγηθούν οι καταναλωτές προς την ε, ε, αγορά καθαρότερων οχημάτων, τότε θα βελτιώσουμε την συνολικότερη κατάσταση αλλά θα χρειαστεί οπωσδήποτε να υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες, αν όχι εναρμονισμένοι, θα πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσει μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να υπάρχει μια ανταλλαγή γνώσεων και να μπορέσουμε από κοινού να οδηγηθούμε ε, μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε και εμείς εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν πάρα πολλές εθνικές αρμοδιότητες ακόμη οι οποίες και ε, προκαλούν το, το φαινόμενο αυτό διαφόρων εθνικών πρωτοβολιών. Καταλαβαίνω ωστόσο ότι αυτό δεν σας βοηθά πάντοτε και ότι ε, πρέπει να σας πω ότι είναι και κάτι ε, δύσκολο να αποφευχθεί στο υπάρχον και ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μπέρς θέλει να μιλήσει, να απαντήσει σε όσα ακούστηκαν. Ναι, παρακαλώ. Γιατί πρέπει να περάσουμε και στις αεροπορικές μεταφορές και στις πλωτές μεταφορές. Ε, δεν αναφερθήκατε καθόλου στις ε, κοινέ μεταφορές, στις συνδυασμένες μεταφορές. Υπάρχουν εμπορικές μεταφορές οι οποίες ε, στα πούλμαν και στα φορτηγά ε, και στα ταξί προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και δεν μιλώ για επιβατικά οχήματα. Μιλούμε για μια μεταστροφή εντός του ίδιου του κλάδου των οδικών μεταφορών. Και να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Η Γερμανία ως αγορά 100, ε, από τα 178.000 ε, λεωφορεία ε, τα 168.000 από αυτά ε, είναι πετρελαιοκίνητα. Αν λοιπόν ε, αλλάξει η σύσταση, τον, ε, η, σύνθεση ε, και μετατρέψεις όλα, το, όλα τα λεωφορεία σε ηλεκτροκίνητα, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση διότι τα λεωφορεία στην πραγματικότητα βοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Πάμε στον κύριο Νοβατσίκ το, από την Airbus Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα. Μιλήσαμε για την αποτελεσματικότητα των κινητήρων και σίγουρα η Airbus ασχολείται με το ζήτημα αυτό καθημερινά. Ξέρουμε ότι γίνεται όλο και καλύτερη η απόδοση, αλλά υπάρχουν κάποια όρια. Ποια άλλη στρατηγική λοιπόν αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Airbus για να μειώσει τις εκπομπές ε, που φυσικά μεταφράζονται και σε ενεργειακό κόστος, σε σημαντικό κίνητρο για τους αερομεταφορείς. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Συντονιστή, ευχαριστώ που με καλέσατε να μοιραστώ κάποιες ιδέες μαζί σας για την κριτικότητα χαμηλών εκπομπών. Να ξεκινήσω με τα καλά νέα. Όλα τα απαραίτητα θεμέλια για τη μείωση των εκπομπών έχουν εντοπιστεί, αλλά ορισμένα θα χρειαστούν ειδικότερη προσοχή. Όπως είπατε, το μεγαλύτερο επίτευγμα προέρχεται από τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των Airbus. Το τελευταίο Airbus, το Α350, έχει 80% καλύτερη απόδοση από το πρώτο αεροσκάφος που υπήρξε. Ε, ε, το όραμά μας είναι μέχρι το 2050 75% μείωση των καυσίμων. και υπάρχει η Project Team Sky ως ε, πλατφόρμα για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Σε παγκόσμιο εμπόδιο, ε, επίπεδο η ΚΑΟ πρόσφατα υιοθέτησε ε, πρώτα μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων ε, που θα ξεκινήσουν από το 2020. Ένα άλλο σημαντικό θεμέλιο λήθος είναι ο τρόπος ε, με τον οποίο διαχειριζόμαστε την ε, ενέργεια κυκλοφορία. Πόσο γρήγορα ουσιαστικά, πόσο μακριά και πόσο αποτελεσματικά πετάνε τα αεροπλάνα. Ε, προς το παρόν χρησιμοποιούνται αεροδιάδρομοι οι οποίοι είναι μακρύτεροι, καθιστούν τα ταξίδια μακρύτερα. Με τις νέες τεχνολογίες θα γίνουν όλα πιο αποτελεσματικά και κατά την άνοδο και κατά την κάθοδο και κατά την πλοήγηση. Μπορεί έτσι να μειωθεί η εκπομπή ε, καυσαερίων ε, κατά 10%. Πέραν όλων αυτών έχουμε άλλο ένα το μέτρο καθώς μιλάμε για ηλεκτροκίνηση και υβριδικά Έχουμε και τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα που θα παίξουν ζωτικό ρόλο στο να επιτύχουμε τους μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Η αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας που θα ζητηθεί σύντομα εδώ αποτελεί ευκαιρία να οριστούν οι συνθήκες της αγοράς που θα δώσουν τη δυνατότητα παραγωγής εναλλακτικού καυσίμου για τα αεροπλάνα που θα δημιουργήσει οικονομικό φύλλο στην Ευρώπη και θα έχει βιωσιμότητα. Το τελευταίο που ήθελα να πω αφορά την πρόσφατη συμφωνία της ΣΥΚΑΟ πρώτο παγκόσμιο σύστημα αντιστάθμιση άνθρακα για την αεροπορία, πρέπει να καταλάβουμε ότι η αύξηση των εκπομπών ε, το, από την αεροπορία οφείλεται κυρίως ε, ε, σε αεροσκάφη εκτό Ευρωπαϊκής Ένωση. Οπότε είναι σημαντικό να εμπλέξουμε και χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πρέπει εμεί να επιδιώξουμε την ανάπτυξη αυτού του θεμελιού υπερασπίζοντας την συμμετοχή τρίτων χωρών ε, στο σύστημα αυτό, αλλά και ε, χρησιμοποιώντας κοινοποιώντας τις τρίτες χώρες ε, μέσω εκπαίδευσης τα δικά μας συστήματα εξοικονόμησης. Θα πρέπει να αποφεύγουμε λοιπόν το διπλό υπολογισμό και να επιδιώξουμε διοικητική απόδοση. Οπότε κάνουμε έκκληση σε εσά να δράσετε για να βελτιώσουμε αυτούς τους θεμέλιους λήθους ε, που απαιτούν ένα πρακτικό ε, νομοθετικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και τα οικονομικά κέρδη του τομέα στην Ευρώπη. Uh, υπάρχει ένα πακέτο μέτρων που συζητεί στην τομέα των αερομεταφορών. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με τα εναλλακτικά καύσιμα. Ε, Βεβαίω υπάρχει αποτελεσματικότητα, αλλά τα εναλλακτικά καύσιμα αργότερα λέτε η τεχνολογική ουδετερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για τους πολιτικούς θύμιτες αφενός. Από την άλλη, όταν μιλάμε για βιοκαύσιμα, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τεχνολογική ουδετερότητα, οπότε πώς θα τετραγωνίσετε τον κύκλο εδώ, διότι αν δείτε τη συζήτηση που γίνεται για την οδηγία για τα ανανεώσιμα, δεν υπάρχει εκεί τεχνολογική ουδετερότητα σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα, διότι ε, τα προωθούμε, τα προωθούμε συγκεκριμένα. Οπότε, το ερώτημα μου είναι το εξή εάν εμείνουμε στην τεχνολογική ουδετερότητα, πώς πιστεύετε ότι τα εναλλακτικά καύσιμα στον τομέα των αερομεταφορών θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν. Βεβαίω ε, μπορεί να γίνει αυτό χωρίς συγκεκριμένη τεχνολογική πολιτική. Είναι και αυτό μια δυνατότητα. Ναι, εξαρτάται τι εννοείται όταν μιλάτε για τεχνολογική ουδετερότητα. τα αναλλατικά καύσιμα είναι τα βιοκαύσιμα όντως, αλλά δεν είναι μόνο. Αυτό δεν γίνεται μόνο μέσω βιομάζας. Υπάρχουν καύσιμα τα παίρνουν ουδέτερα για τις αεροσκάφη. Ε, όπου δεν αλλάζει δηλαδή κάτι στην κινητήρα. Αλλά υπάρχει ε, και το θέμα του τύπου των ε, ε ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται. Υπάρχει ένας κατάλογος σχετικός. Πρέπει στο μέτρο του δυνατού βεβαίως να είμαστε ουδέτεροι, διότι δεν υπάρχει ε, καλό και κακό ε, καύσιμο, υπάρχει ε, καλή και κακή πρακτική. Αυτό που λείπει για την ώρα στην ευρωπαϊκή πολιτική είναι ένα σαφές κριτήριο βιωσιμότητας. Υπάρχει περιθώριο ε, καινοτομίας, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, την καινοτομία με τόσους περιορισμούς και βεβαίως υπάρχει το θέμα των συνθήκων της αγοράς. Η πραγματικότητα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των καυσίμων που εισάγονται στην Ευρώπη, βιοκαυσίμων εννοώ, ε, δεν πάνε στον τομέα των αερομεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες στην αγορά έτσι ώστε ο τομέα, ο αεροπορικό, να αγοράζει τα καύσιμα και να δημιουργήσουμε και τι συνθήκε στην αγορά για να παράγουμε αυτά τα βιοκαύσιμα στην Ευρώπη. Και έχουμε, έχουμε γι' αυτό υπάρχει προτήλη, διότι έχουμε τα, ε, βιοαπο, τα ε, Και τώρα να περάσουμε στο νερό, στους υδάτινους ε, στις θαλάσσιες οδούς, τις εσωτερικές ε, οδούς, συγγνώμη. Ε, μιλάμε για συνδυασμένες μεταφορές, ε, οδικές, σιδηροδρομικές και, και εκεί στις συνδυασμένες μεταφορές μπαίνει και το θέμα των εσωτερικών ε, πλωτών οδών. Ο κλάδος σας ποια θέση έχει σε αυτό το σύστημα και πώς το, τι μεταχείριση τη από τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ κύριε Εκχάουτ, καλημέρα. κύριε και κύριοι, Όταν μιλάμε για μεταφορές ε, μεγάλων αποστάσεων, ε, συνήθως ε, έχουμε, μιλάμε για κάποια μεγάλα πλοία που κουβαλάνε χημικά απόβλητα, χημικά προϊόντα ή κατασκευαστικά υλικά ε, και αυτά γίνονται όπου, υπάρχει μια καλή, όπου υπάρχουν υποδομές καλής ποιότητας. Ε, στον διάδρομο των, ε, του Ρήνου και των Άλπεων, ε, ως ένα βαθμό και στο Δούναβι, σε κάποιους άλλους ακόμα οδούς. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα κοντέινερ, τα οποία ακολουθούν τις ίδιες, ε, τις ίδιες πλωτές οδούς. εκεί υπάρχει βεβαίως ανταγωνισμός, φυσιολογικό αυτό. Θα θέλαμε όμως ίσε ευκαιρίες, ίση μεταχείριση. Όταν υπάρχουν δηλαδή επιδοτήσει σε ένα κλάδο θα θέλαμε ε, αυτές οι επιδοτήσεις να πάνε και σε άλλους κλάδους ε, ή αλλιώ να μην υπάρχουν καθόλου επιδοτήσει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ε, πού βλέπετε να υπάρχουν επιδοτήσεις ε, και, να, και πού να μην υπάρχουν, διότι το είπατε κάπω γενικά, μπορείτε να γίνετε κάπω πιο συγκεκριμένοι. Ναι, ακούστε, στον τομέα της πλοήγησης βεβαίως υπάρχει ο ανταγωνισμός ε, που έχει να κάνει με το επίπεδο του ύδατος, αν έχουμε χαμηλό επίπεδο ύδατος, τότε αναζητώνται εναλλακτικέ λύσεις, λογικό αυτό ε, και επιθυμητό. Ε, έτσι έχουμε τις συνδυασμένες υπηρεσίες, υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών. Τώρα, σε κάποιες χώρες όμως υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης για συγκεκριμένες μεταφορές, για να μεταφερθούν, παραδείγματος χάρη, κάποια ε, υλικά με ένα συγκεκριμένο τρόπο μεταφοράς και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για τους υπόλοιπους. Ε, υπάρχει και ανταγωνισμός ε, μεταξύ των, των διαφορών τρόπων μεταφοράς. Στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, ε, χρησιμοποιούνται συχνά αυτές οι πρωτές οδούς, διότι υπάρχει νερό παντού Επίσης είναι τόσο υψηλό το κόστος ε, ε για τους ε, ε, για τους πιλότους είναι πολύ υψηλό ε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα ανταγωνισμού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τις ευκαιρίες για όλους για να είναι το ίδιο εύκολο να επιλέγει κάποιος μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Να επιλέγει ο καθένας αυτό που τον βολεύει καλύτερα, αυτό που του ταιριάζει καλύτερα, να υπάρχει ουδετερότητα. Ε, τώρα, ε, όταν σκεφτόμαστε για πλωτές οδούς, ε, συνήθως ε, θεωρούμε ότι μιλάμε για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, αλλά οι αποστάσεις μειώνονται. Μειώνονται διότι υπάρχει σημαντική επένδυση και εδώ μιλάω βέβαια για την οργάνωση να οποία εκπροσωπώ, διότι εμεί ασχολούμαστε, είμαστε διαχειριστέ πλωτών οδών μεταφορών ε, ε, γίνονται λοιπόν πολλές επενδύσεις ε, στην υπηρετική μεταφορά, στην αστική μεταφορά και βεβαίως έχουμε κάποια πάρκα, παραδείγματος χάρη οικοβιομηχανικά και εκεί πια είναι μικρές οι αποστάσεις. Και όταν μιλάμε για εκπομπές και εδώ είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουμε σε ηλεκτρονική ενέργεια, για τις μεγάλες αποστάσεις είναι πιο δύσκολο εκεί εξετάζουμε το LNG, αλλά ε, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε και το diesel όσο γίνεται περισσότερο και βέβαια diesel με όσο γίνεται με μικρότερο, ε, μικρότερη ποσότητα εκπομπών. Για να φτάσουμε βέβαια σε μηδενικές εκπομπές, αυτό είναι ακόμα δύσκολη πρόκληση για μας. Χρειάζεται έρευνα, ε, έρευνα και με τις θαλάσσιες μεταφορές βεβαίως, αλλά αλλά ε, δεν είναι πάντα το ίδιο. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται στους αλλάξεις τομέας δεν είναι ο ίδιος με αυτά που χρειάζεται το τομέα των πλωτών εσωτερικών οδών, οπότε δεν πρέπει να το συνδυάζουμε απαραίτητα σε έρευνα. Έχουμε ακόμα λοιπόν δουλειά μπροστά μας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στον τομέα των εκπομπών είναι βεβαίως, ε, και εδώ συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές, δεν είναι μόνο ε, θέμα ε, στοιχείων ε, για τις καθημερινές εκπομπές. Ε, ξέρετε ότι ορισμένε φορές ορισμένα πλοία είναι ηλικιωμένα, είναι παλιά, μπορεί να έχουν νέους κινητήρες, αλλά δεν αναμένουμε ε, τα πάντα από αυτά τα νέα πλοία, διότι και η κατασκευή νέων πλοίων παράγει εκπομπές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα ε, να ε, διαχειριστούμε αυτά τα πλοία για να μπορέσουν να, να κρατήσουν για πιο πολύ καιρό. Ναι, είδατε ότι είναι χαμηλότερο το κόστος σε αφορά τους εθνικούς πρώτες οδούς, αλλά ήταν υψηλή η μόλυνση της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει να κάνει με τον δίζελ προφανώς. Αναφερθήκατε ήδη βέβαια σχετικά. Ε, πώς πάνε οι επενδύσεις ε, έτσι ώστε αυτό το εξωτερικό κόστος να μπορέσει να μειωθεί. Ποιες είναι οι προοπτικές για να μειωθεί αυτό το κόστος συγκεκριμένα. Ναι, ακούστε, υπάρχουν πολλές και διάφορες. Το πιο απλό, ας πούμε, είναι η επεξεργασία εκ των υστέρων. Έχουμε, να έχουμε καταλύτες δηλαδή, να έχουμε φίλτρα σε ό,τι αφορά τα σωματίδια ε, και είναι και το πιο, πιο φθηνός τρόπος αυτός. Από εκεί και πέρα μπορεί να, να αλλάξουμε, να βρούμε άλλους τρόπους ε, όθησης. Ε, υπάρχει αυτό ήδη, αλλά για πιο μικρά, μικρές οδούς, ε, ε, για πιο σύντομες οδούς. Και εκεί βεβαίως πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Έχουμε και το LNG, αλλά και εκεί χρειάζεται επεξεργασία εκ των υστέρων για να είναι όσο γίνεται μικρότερες εκπομπές. Ε, η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε εκεί είναι το κόστος. Και αυτό που θα θέλαμε πραγματικά να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι εδώ είναι η μοιρασμένη ευθύνη από πλευρά των ρυθμιστικών αρχών αλλά και από πλευρά των καταναλωτών. Ε, η καινοτομία πρέπει να επιβραβεύεται. Ε, αυτή τη στιγμή όταν κάποιος επενδύει σε ένα νέο σε μια νέα μορφή κινητήρα, σε ένα νέο κινητήρα ε, και βεβαίως θα βρεθεί με χρέη και δεν είναι βέβαιο ότι θα τον επιβραβεύσει ο πελάτης και αυτό είναι κακό για τον ανταγωνισμό. Και αν κάποιο θέλει να περάσει το υδρογόνο, παραδείγματο χάρη, ε, ε, δεν μπορεί ε, να θέσει ένα τέτοιο πλοίο σε εμπορία, διότι το επιτρέπει ο κανονισμό. Και εκεί λοιπόν θα χρειαζόμαστε ε, μεγαλύτερη ευελιξία σε κανονιστικό επίπεδο για να μπορούν να επιτρέπουν τέτοιου καινοτομίε. Μάλιστα, το λάβαμε το μήνυμα. Να περάσουμε τώρα στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Βεούβεν. Το πιο απλό ερώτημα είναι η εξελίξη των τομέων θαλάσσιων μεταφορών. Ποιε είναι οι προσδοκίες για τεχνολογική πρόοδο για να μειωθούν οι εκπομπές και βεβαίως βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Τι αναμένεται και πόσο γρήγορα θα πάμε εκεί. Καλησπέρα. Ναι, υπάρχουν πράγματι πολλές εξελίξεις που πρέπει να τις ε, εξετάσουμε προσεκτικά και ξέρετε ότι τα μέτρα που αναπτύσσονται για, τις, ε, για την αυτιλία ε, ε, αναπτύσσονται σε επίπεδο IMO με βασικότερο στόχο την ε, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας με προδιαγραφές και πρότυπα τόσο για τα νέα πλοία όσο και για τα υπάρχοντα πλοία. Εξετάζοντας λοιπόν το μέλλον και τις επιπτώσεις που θα έχουμε, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, δηλαδή τις εκπομπές ανά χιλιόμετρο, περιμένουμε ε, μια μείωση 50% έως το 2050. Αυτό βέβαια είναι σχετικό. Άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι ε, πώς θα ε, προχωρήσουμε με την απόλυτη μείωση των εκπομπών. Αυτό σχετίζεται και με το ευρύτερο πλαίσιο των στόχων του Παρισίου και την στρατηγική που θα εκπονήσουμε ως IMO τις επόμενες, το, επόμενο διάστημα, για τις επόμενες δεκαετίες. Και φυσικά είναι σαφές ότι ε, θα εξακολουθήσουμε για αρκετό καιρό ακόμα να εξαρτώμαστε από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε ε, μια σοβαρή εναλλακτική η οποία να μπορεί να ε, αναπτυχθεί και να επεκταθεί στο 100%. Εξετάζουμε διάφορες ε, εναλλακτικές, υδρογόνο, μεθάνιο ε, τα λοιπά Αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάποια εναλλακτική λύση η οποία να μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τα επόμενα 20-30 χρόνια σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε από ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και άλλους ε, μηχανισμούς ώστε να καταφέρουμε ως κλάδος να επιτύχουμε τους στόχους του Παρσίου Και αυτή είναι, είναι η ουσία που θα έχουμε ε, στο πλαίσιο του, της συζήτησης που θα έχουμε έως το 2018 ε, στον IMO. Ε, μιλούμε δηλαδή για τις προδιαγραφές για τα νέα πλοία, για, τα, για τις προδιαγραφές για τα υπάρχοντα πλοία, αλλά και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο μεσοδιάστημα αλλά βεβαίως και πώς μπορούμε να προωθήσουμε την έρευνα, την ε, καινοτομία ώστε να εξασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε την ε, ε, απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη και την επέκταση νέων μορφών τεχνολογίας. Αυτή θα είναι η συζήτηση που θα έχουμε στο πλαίσιο της στρατηγικής του IMO τα επόμενα δύο χρόνια. Μια ακόμη ερώτηση και μετά θα σταματήσω. Σε ποιο βαθμό χρειάζεστε ε, τη βοήθεια των φορέων χάραξης πολιτικής. Ξέρω ότι ο ΑΕΜΟ εσωτερικά κάνει αυτή τη συζήτηση, την παρακολουθούμε, όμως τι, χρειάζεται, τι χρειάζεστε από τη σκοπιά του πλαισίου πολιτικής προκειμένου να ε, διευκολυνθεί και η συζήτηση που εσείς κάνετε. Αν δούμε την ευρωπαϊκή πολιτική συγκεκριμένα, προφανώς χρειαζόμαστε τη συμβολή και την ε, ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι ο IMO αποτελείται από 177 μέλη. Πολλά μέλη του είναι ε, ε, ευρωπαϊκές χώρες. Χρειαζόμαστε και τη δική τους συμμετοχή και συμβολή ώστε να μπορέσουμε να, να φτάσουμε και να απευθυνθούμε και ενδεχομένως και σε άλλους εταίρους, μέλη του IMO, οι οποίοι πιθανόν να είναι λιγότερο φιλόδοξοι ως προς τους στόχους τους. Δεύτερον, χρειαζόμαστε υποστήριξη για την καινοτομία, ε, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Έχουμε ήδη μια σειρά από μέσα και εργαλεία, το TNT, το ΣΕΦ, υπάρχουν ε, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, αυτόν τον, αυτε, του, αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες πράγματι βοηθούν από την Ευρώπη και νομίζω ότι ε, μπορούν να τροφοδοτήσουν με θετικό τρόπο και τη στρατηγική που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, υποστήριξη ε, στο τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και υποστήριξη στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το, αυτή τη χρονοθυρίδα, αυτό το χρονοδιάγραμμα έως το 2018 με, που θα γίνει η κατάρτιση, η οριστικοποίηση της στρατηγικής του IMO ε, και στο, στην κατεύθυνση αυτή θα χρειαστούμε την βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για να αποκτήσουμε μια εποπτεία επί των διαφόρων ε, τρόπων μεταφορών που υπάρχουν. Φυσικά είναι αδύνατο να καλύψουμε όλα τα θέματα μέσα σε 45 λεπτά. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστούμε γιατί νομίζω ότι σχηματίσαμε μια καλή εικόνα. Ακούσαμε και ορισμένες επιθυμίες και ε, ορισμένα αιτήματα των ε, κλάδων και θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Πρόεδρο ώστε να συνεχίσουμε με την συνεδρίασή μας. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στους συντονιστές μας οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες, εκπροσωπούν όλους τους τομείς ε, και τους κλάδους. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε ερωτήσεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Βιμ Βαντερμπροκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Εγώ μιλάω στα Ολλανδικά αφού υπάρχουν ένα σωρό συμπατριώτες μου και φίλοι Φλαμανδοί. Έτσι λοιπόν να ασκηθούμε και λίγο. Λοιπόν, πρώτα πολλά να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου μα Εμιλιανό Σαλίνη, ο οποίο ε, είχε μια υποχρέωση τελευταία στιγμή ε, στη ε, Ρώμη και είναι και ο σκιώδης για την έκθεση του Μπας Eichhout εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Θα θελήσει λοιπόν να ενημερωθεί για αυτή τη συζήτηση. Έχω πέντε ερωτήσεις, αλλά να κάνω μια εισαγωγή για να εξηγήσω τη θέση του ΕΛΚ με δύο-τρία λόγια. Λοιπόν, το ΕΛΚ ως ομάδα θέλει να διατηρηθεί η έννοια των διατροπικότητα. διατροπικότητας. Δεν θέλουμε να τιμωρηθεί ο, ο δικός κλάδος, θέλουμε να βελτιωθεί. Είναι λοιπόν διαφορετική η προσέγγιση μα γιατί άλλες ε, πολιτικές ομάδες θέλουν να τον καταργήσουν. Εμείς απλά θέλουμε να τον βελτιώσουμε, να το καταστήσουμε πιο ε, εξειδικευμένο. Εγώ στην εσωτερική ομάδα, του, εντός της ομάδας του ΕΛΚΑ, ασχολούμαι με τις ε, δραστηριο... συγκεκριμένες δραστηριότητες μεταφορών που αφορούν τις οδικές και τις διατροπικές. Όταν μιλάμε για περισσότερη βιωσιμότητα όμως, πρέπει να δίνουμε και κάποια νούμερα. Τα νούμερα αυτά δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2015 και το ΕΛΚ θέλει να βασιστεί σε αυτά τα στοιχεία για τη συνεργασία. Διακρίνουμε κάποια αισιοδοξία, υπάρχει μια ελπίδα να επιτευχθούν οι στόχοι και υπάρχει και κάποιος ρεαλισμός ε, μεταξύ καταναλωτών, παραγωγών Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφιλειώσουμε και τις δύο αυτές ε, θέσεις, διότι μαζί με τον εισηγητή δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του Συμβουλίου. Θα πρέπει να σκεφτούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ αισιοδοξία και ρεαλισμού. Να μην πέσουμε στην παγίδα του Συμβουλίου, διότι διαφορετικά θα αρχίσουν να εκφράζονται πολλά εθνικά συμφέροντα σε αυτές τις πολύ δύσκολες πολιτικές εποχές. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον εκπρόσωπο των Ελβετικών Σιδηροδρόμων, τον, ή μάλλον τον κύριο Σούτερ, γιατί υπάρχουν ναι, αυτές οι δαπάνες, οι εξωτερικευμένες δαπάνες των 510 δις. Εδώ και χρόνια μελετάει η Κομισιόν αυτό το φάκελο. Πώς καταλήγεται σε αυτό το νούμερο. Εγώ σε επαφές μου με την Κομισιόν ε, έμαθα ότι πρέπει να περιμένουμε το 2018 δύο νέες μελέτες. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Ζωνάρα. Πρόσφατα μάθαμε νέα κριτήρια για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Daimler Mercedes, η Volkswagen υλοποιούν τα κριτήρια αυτά ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο στην Ευρώπη. Μετά μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ερμπάς όπου μάλιστα είχαμε και μια πρόσφατη επίσκεψη και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη για μας. Μιλήσαμε για στόχους εκπομπών για το 2050. των εκπομπών των αερομεταφορών. Ε, μιλάμε για σημαντικές ε, ε, ε, μειώσεις μέχρι το 2050. Εδώ θα πρέπει να εκφράσουμε κάποιο ρεαλισμό και κάποια αισιοδοξία και όλα θα βασιστούν στην τεχνολογία. Ε, τώρα για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Εμείς δυστυχώς εδώ βρισκόμαστε ενώπιον παλιών φορτηγίδων με ε, κινητήρε 30 ετών είναι απερχαιωμένοι και σε περίπτωση που καταρρεύσει η αγορά θυμάστε το 2009 η αγορά βρέθηκε σε πολύ αδύναμη θέση τι έπρεπε να κάνουμε να αντικαθιστούμε ταχύτερα τους κινητήρες των φορτηγίδων ε, και μετά μία ερώτηση προς τον κύριο Φερχόβεν. λήφθη η απόφαση για το ETS ε, για το 2025 η οποία θα εφαρμοστεί ήδη από το 2023 όπως μας είπε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας. Συγγνώμη, όλα αυτά ε, δεν, το δεν τα ποικοτάρουν κάπως οι Κινέζοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αρτούγκ. Ευχαριστώ πολύ τους ε, πυρογνώμονες για τις παρουσιάσεις τους. Νομίζω ότι ε, επανερχόμαστε πολύ συχνά στα ίδια και στα ίδια θέματα. Και πλέον οι εκπρόσωποι των ε, διαφόρων κλάδων έχουν εκθέσει τις απόψεις τους και γνωρίζουν πλέον και οι ίδιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανάγκη επιτέλους να υποβάλει μια ε, γενική έκθεση ώστε να έχουμε εικόνα για το πόσο ο κάθε τρόπος μεταφορών τελικά συμβάλλει ε, στις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ε, καλό ε, είναι να γνωρίζουμε ποιος τελικά ρηπαίνει και ποιος πληρώνει, διότι αλλιώς έχουμε αυτό το διαρκές γαϊτανάκι αλληλοκατηγοριών ότι ναι εμείς πληρώνουμε όμως ήδη πάρα πολύ κτλ. κτλ. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο είναι η Κομισιόν να συντάξει μια γενική έκθεση επισκόπησης ώστε να συγκεραστούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε και εμείς να ε, εξαγάγουμε τα ενδεδειγμένα συμπεράσματα. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε την κατάσταση κατά την οποία κάθε επιμέρους ε, τρόπος μεταφοράς κάνει για τον, για τον εαυτό του ε, έρευνες και δίνει τα στοιχεία του. Ε, αυτό όμως δεν μας βοηθά να προχωρήσουμε. Ε, ελπίζω ότι η συζήτηση δεν θα είναι η ίδια αυτή τη φορά με εκείνη που είχαμε πριν από 10 χρόνια όπου ε, συζητούσαμε στην ουσία ακριβώς τα ίδια θέματα και τελικά καταλήξαμε σε έναν συμβιβασμό. Θα ήταν πάρα πολύ κρίμα να μην επιτύχουμε παρά την πάροδο 10 ετών να μην καταλήξουμε σε τίποτα ουσιώδες. Άρα, ε, να ξεκινήσουμε από μια τάμπουλα ράσα, να μας πει η Κομισιόν τι ακριβώς συμβαίνει, να δούμε ποιες είναι οι επιβαρύνσεις, οι περιβαλλοντικές, σε 28 κράτη-μέλη, διότι φυσικά η αεροπορία, για παράδειγμα, στην Γερμανία επιβαρύνει με διαφορετικό τρόπο το περιβάλλον στη Γερμανία από ό,τι σε άλλες χώρες. Οι οδικές μεταφορές έχουν διαφορετικό μερίδιο ε, συνεισφοράς στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, στη Γερμανία από ό,τι ενδεχομένω σε άλλες ε, χώρες. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και μια, υπάρχει και μια πλειάδα μέτρων τα οποία λαμβάνονται όπως είναι για παράδειγμα τα Γερμανία που εισήχθησαν πρόσφατα τα διόδια που εισήχθησαν πρόσφατα στη Γερμανία χωρίς ωστόσο να υπάρχει συντονισμός και εναρμόνιση Άρα αυτό που μπορώ να κάνω εγώ από την πλευρά μου είναι άλλη μια φορά να απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν επιτέλους να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία και να υποβάλει μια γενική έκθεση γιατί αλλιώς θα έρθουμε και σε 10 χρόνια και πάλι θα συζητούμε για τα ίδια θέματα. Και τώρα η άλλη συντονίστριά μας, η κυρία Κίλωνεν, για την ΚΟΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τους πελάτες. Οι πολίτες έχουν πολλά ερωτηματικά. Ταυτόχρονα. Η παραγωγή των εκπομπών, κλιματική αλλαγή, αποδοτική χρήση της ενέργειας, κυκλική οικονομία, φορολόγηση, συστήματα πληρωμών, καύσιμα και νέα καύσιμα, νέες τεχνολογίες, η προώθησή τους. Πώς λοιπόν μέσα σε όλο αυτόν τον κικαιώνα μπορούμε ή μπορούν οι συμπολίτε μας, οι καταναλωτές να συμμετέχουν συμμετέχουν, να παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές. Διότι προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι και οι προσωπικές επιλογές επηρεάζουν, επιδρούν πάνω στα ζητήματα αυτά. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος δεν έχει χρήματα είναι πολύ δύσκολο να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, να προωθήσει ε, το οτιδήποτε με την ε, συμπεριφορά του. Ε, ακόμα και η προσπάθεια που γίνεται για να αποτραπεί η κλιματική αλλαγή. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πώς θα κάνουμε σωστές αναλύσεις κόστους που θα μας βοηθήσουν εμάς ως πολιτικούς συνήθες αλλά και τον κλάδο ή και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους κλάδους Πώς θα μας βοηθήσουν λοιπόν τα στοιχεία αυτά ε, να κάνουμε τις σωστές, τις έξυπνες επιλογές οι οποίες ταυτόχρονα ε, θα μειώσουν ε, βεβαίως τις ε, βλαβερές εκπομπές αλλά δεν θα οδηγούν σε μια κατάσταση όπου δεν θα είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση περιβαλλοντικά. Μάλιστα, παρακαλώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Λούντγκρεν. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ε, αφέλεια στη συζήτηση αυτή. Αν δούμε τι γίνεται στον, ε, στις οδικές μεταφορές, παραδείγματος χάρη, κάποιοι λένε ότι είναι λύση για το μέλλον αυτό ε, με τα λεωφορεία που κυκλοφορούν πάνω σε τρένα. Ακούστε, ε, στο 90% των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται λεωφορεία, παραδείγματο χάρη. Ε, των φορών που χρησιμοποιούνται λεωφορεία έχουμε 1,6 ε, επιβάτες. Οπότε για να είναι περιβαλλοντικά φιλικό προ το χρήστη πρέπει να είναι 90 επιβάτε για να είναι όσο φιλικό προ το χρήστη είναι το να κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο με ένα άτομο. Ένα λεωφορείο καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα ε, δεν μπορεί να είναι 100% πλήρε, όπω αντιλαμβάνεστε ίσως σε μια μεγάλη πόλη. Αλλά μόλι βγούμε από τι μεγάλου πόλει, τότε ε, έχουμε πολλά λεωφορεία ε, εντός των οποίων είναι λίγοι επιβάτε και κοστίζουν ή μάλλον δημιουργούν περισσότερες εκπομπές από ότι τα ΙΟΤΑΧΗ και το ίδιο ισχύει και με τα φορτηγά. Όταν το χρησιμοποιεί κάποιος στο Παρίσι, ε, οι εκπομπές που υπάρχουν είναι βεβαίως πιο καθαρές από αυτήν ε, από τον αέρα, την ατμόσφαιρα ε, στην Γαλλία, ε, στο Παρίσι, όπως περιπτώσει. Στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, υπάρχει μια νομοθεσία, τουλάχιστον μας δω την κατάσταση στη Σουηδία, εκεί βλέπουμε ότι η νομοθεσία επιτρέπει έχουμε τεχνολογία 20 ετών από τις πρώην ανατολικές χώρες. Και βεβαίως πολλοί χρησιμοποιούν το ντίζελ από τις ανατολικές χώρες. Έρχονται αυτά τα οχήματα στη Σουηδία και εκεί, όπου πρέπει, εκεί πρέπει να χρησιμοποιείται ντίζελ περιβαλλοντικής κλάσης 1. Όμως είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε αλλοδαπούς ε, ε, οδηγούς που έρχονται στη δική μου χώρα ε, και μολύνουν την ατμόσφαιρα, στη Σουηδία, με αυτό το βρώμικο ντίζελ. Γιατί το κάνουν αυτό, λόγω της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας τους επιτρέπεται να το κάνουν. Και αν δείτε τώρα τα γιοταχή, τα ηλεκτρικά οχήματα, για μένα αυτό δεν έχει βγάζει κανένα νόημα. Παράγουμε την ενέργεια αλλού. Και βεβαίως ε, σκεφτείτε και τις μπαταρίες που θα χρειαστούν, έτσι. Οι μπαταρίες ε, ε, είναι τοξικά υλικά, είναι ε, δηλητήριο. Τι θα γίνει με τις μπαταρίες όταν τελειώνει ο κύκλος ζωής τους. Λοιπόν, δεν νομίζω αυτή η εναλλακτική να αποτελεί λύση. Πρέπει να βρούμε ενδεχομένω κάποια, νέα, κάποια νέα μορφή καυσίμου. και βεβαίως χρειαζόμαστε κανόνες ε, που να μην επιτρέπουν η Σουηδία αυτή τη στιγμή να πλημμυρίζει από φορτηγά. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε του συντονιστέ. Να δώσω το λόγο σε κάποια μέλη. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, αγαπητοί συναδέλφοι. Έχετε ένα λεπτό για να κάνετε τι ερωτήσει σα. Ε, να είστε πολύ ακριβεί λοιπόν και γρήγοροι. Δίνω το λόγο στην κυρία Λουκασένκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι περίπλοκο το θέμα. Ένα λεπτό είναι σίγουρα λίγο, αλλά η συζήτησή μας δείχνει πόσο δύσκολη είναι, είναι το θέμα. Το να συζητάμε τα αγωνιστικότητα και μείωση των εκπομπών είναι κάτι περίπλοκο. Οπότε τα όνειρά μας, οι αποφάσεις μας, οι συμφωνίες μας, τα σχέδιά μας ε, υπερβαίνουν τις δυνατότητες που έχουμε και σε ορισμένες χώρες δεν είναι καν κοινωνικά αποδεκτές. Ας σας μιλήσω τώρα για την ουσία. Μιλάμε για τα ηλεκτρικά οχήματα. Κατά την άποψή μου, σωστή η κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την υποδομή που απαιτείται. Δηλαδή μπορεί να οδηγήσει κανείς 100 χιλιόμετρα χωρίς να χρειάζεται να φορτίσει την μπαταρία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει κανείς στον αυτοκινητόδρομο. Τώρα όσον αφορά τα βαρέα οχήματα, τα οποία ενδέχεται να πάνε σε κάποιες χώρες, ε, το συζητήσαμε. Δεν έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο να συζητήσουμε για τα βαρέα οχήματα, διότι οι κινητήρες τους δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα τα οποία θα έπρεπε. Ειδικότερα όταν μιλάμε για φορτηγά που έρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται και το θέμα τη ποιότητα του καυσίμου που για παράδειγμα είναι διαφορετικό στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει ψάξει κανένα. Το καύσιμο αυτό επιτρέπεται στη δική μα έννοια αγορά. Και το επόμενο τώρα, ε, οι ε, μεταφορές μας, οι κοινέ μας είναι επιβατισμός. Ε, καλό θέμα αυτό, καλή λύση για τις πόλεις, αλλά στις αγροτικές περιοχές ο κύριος Κράμερ. Ε, εκπροσωπώ τον αναλούνται. Ε, γι' αυτό και έχω το λόγο, το, χρόνο του να μιλήσω ως συντονιστής. Ως ε, Όλοι μιλούν για την εσωτερικεύση του κόστης. Όλοι μιλούν υπέρ της κινητικότητας και των μεταφορών. Αλλά θέλουν απλώς να αλλάξουν τα τεχνολογικά μέσα. Μα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εμάς, στόχος μας είναι και να αλλάξουμε τους τρόπους μεταφορών και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά όχι αν μείνουν τα πάντα όσα έχουν. Ξεκινώ ε, με τις οδικές μεταφορές. Ο δήμαρχος του ε, ε, Μονάχου πριν από 45 λεπτά, χρόνια είχε πει ότι το αυτοκίνητο σκοτώνει τις πόλεις μας. Ακόμη και αν αντεκατασταθούν όλα τα αυτοκίνητα σήμερα με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, δεν πρόκειται να ε, αλλάξει το πρόβλημα των, ε, του μποτιλιαρίσματος, των χαμένων ορών εργασίας, της χαμένης παραγωγικότητας. Το, γι' αυτό και πρέπει να αλλάξουμε συνολικά το, την αντίληψή μας για τις ε, μεταφορές. Αν σκεφτεί κανείς ότι ε, το 90% των διαδρομών που διανύονται με αυτοκίνητα έχουν ε, μήκος 6 χιλιόμετρα και ότι 23 στις 24 ώρες της ημέρας τα περισσότερα αυτοκίνητα μένουν ακινητοποιημένα, αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται μια αλλαγή αντίληψης. Αυτό αφορά το 80-85% ε, των ε, κατοίκων των ε, πόλεων. Η αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα, δεν πληρώνουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρο για την κυριοζήνη. Για ε, κάτι που ε, αναγκάζονται όμως να κάνουν οι σιδηρόδρομοι. Γι' αυτό και έχει υπάρξει αυτή η τεχνητή ε, προώθηση των, ε, των αεροπορικών μεταφορών. Υπάρχουν μέχρι και αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ πόλεων που οι, τα ταξίδια θα διαρκούσαν ε, λιγότερο με σιδηρόδρομο από ότι αν τα κάνεις με το αεροπλάνο, αλλά επειδή το αεροπλάνο είναι πιο ε, φθηνό, πολλοί άνθρωποι ε, καταλήγουν να επιλέγουν αυτή τον, αυτόν τον τρόπο. Δεν το λόγο στον κύριο Τεμές Μάκερ. Θα μιλήσω και εγώ Ολλανδικά, με μεγάλη μου χαρά. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Γκέιναρτ. Τον κύριο Ζωνάρο. Ήθελα να μιλήσω για τον στόλο των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανανεώσουμε μια σειρά από κίνητρα φορολογικά. Στη χώρα μου, στο Βέλγιο, υπάρχει ένα σύστημα φορολογικό που δίνει κίνητρα για να χρησιμοποιεί κάποιο τα αυτοκίνητα τα επαγγελματικά των επιχειρήσεων, δηλαδή που οποίε δουλεύουν. Και αυτό οδηγεί στο να υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα βέβαια ε, στο Βέλγιο και πολλοί επιλέγουν να, το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο της δουλειά τους. Και αυτό είναι ει βάρο άλλων μέσων μεταφοράς. Οπότε δεν επενδύουμε σε, άλλες, ε, σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Αυτό έχει επιπτώσει το κόστος, και τα και τα Τώρα, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνεται η εντύπωση ότι διαφέρουν οι κανόνες. Στις μη κοινωτικέ αγορές υπάρχει ένα σύστημα διπλωμάτων βεριστεχνίας διαφορετικό. χρησιμοποιούν δηλαδή άλλες εναλλακτικές που έχουν να κάνουν την εσωτερική καύση. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται συνειδητά από τον κλάδο. Να, επενδύουν, να μην επενδύουν σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία ενώ όλοι οι άλλοι το κάνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ παρακαλώ που προσπαθήστε να είστε σύντομοι γιατί θέλω να έχουμε και απαντήσεις από τους εμπειρογνώμονες. Παρακαλώ. Ε, εντάξει, Λοιπόν, ακούστηκαν πολλά, γνωρίζουμε πολύ ε, ότι ε, βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες πρωτοβουλίες για την μείωση των εκπομπών. Για μένα ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι οι υποδομές για τις εναλλακτικέ μορφές ενέργειας. Είχαμε πριν από δύο χρόνια ε, θεσπίσει ένα νομοθέτημα και θυμάμαι ότι ως κοινοβούλιο είχαμε, θέλαμε μάλλον πολύ πιο φιλόδοξους στόχους ως προς τον, τις ε, χρονολογίες επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα όσα τελικά αποδέχθηκαν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Ε, είχαμε πει τότε να μπορεί κανείς να φορτίζει το, ε, το αυτοκίνητό του ε, σε πολύ περισσότερα μέρη από ό,τι προβλέπετε τώρα. Τώρα, τέθηκε ένα ζήτημα σχετικά με, με το modal shift, δηλαδή την μετάβαση στους τρόπους μεταφορών. Δυστυχώς ε, η συζήτηση επικεντρώνεται πολύ ε, στην ε, μετάβαση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και όχι τόσο στη μετάβαση από τις οδικές στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Δεύτερον, στους σιδηροδρόμους. Αυτό ίσως απευθύνεται στον Ελβετό εκπρόσωπο. Ε, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες έχω την εντύπωση ε, ε, ότι δεν επενδύονται αρκετά χρήματα ώστε να προμηθευτούν οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί τεχνολογίες για την φόρτωση μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και τη μεταφορά τους από τα φορτηγά στους σιδηροδρόμους. Είπατε ότι το, το υδρογόνο ως ε, καύσιμο δεν επιτρέπεται. Ε, το απευθύνω στον εκπρόσωπο ε, του IMO. Να ρωτήσω και ένα, κάτι τελευταίο. Έχετε έναν κατάλογο των χωρών που δεν έχουν ακόμη νομοθετικό πλαίσιο για την ε, ρύθμιση του, του, των, ε, των διατάξεων που διέπουν το, το διοξίδιο του αζότου. Έχετε ε, ίσως ένα κατάλογο των λιμανιών που θα, χρειάζ, που θα χρειαστούν μετασκευή προκειμένου να ανταποκριθούν στις ε, απαιτήσεις της νομοθεσίας. Λοιπόν, έχετε ένα λεπτό, θα σας, κόβω το, θα το μικρόφωνο μετά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να υπάρξουν και απαντήσεις από τους πυρογνώμονες στα όλα αυτά τα ερωτήματα. Κύρια λόγο. Θα προσπαθήσω να τα πω σύντομα. Χρειάζονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Είναι ε, γεγονός ότι ε, οι προθέσεις είναι καλές, αλλά χρειάζομαστε πράξεις. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον ε, βελβετό ε, ε, εκπρόσωπο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτεθεί αυτός ο στόχος του, των 65.000 ε, οχημάτων κατ' έτος στις οδικές μεταφορές. Θέλω να μου πείτε, ε, επειδή εγώ προέρχομαι από το Τυρόλο και από το Μπρένερ περνούν 2 εκατομμύρια φορτηγά κάθε χρόνο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς αυτή τη μετάβαση από τις οδικές στις συνδρομικές μεταφορές. Ε, πώς μπορούμε επίσης να καταστήσουμε πιο κερδοφόρες, επικερδείς τις ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πώς, ποια μέτρα χρειάζονται, θεωρείτε εσείς, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη μετάβαση από τις οδικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να απογοητεύσω τους υπόλοιπους συναδέλφους, οπότε θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Μα έχετε οργανώσει ολόκληρη ομάδα σήμερα το απόγευμα, λέει η Πρόεδρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε όλοι εδώ, απευθύνουμε στου εμπειρογνώμονε. Κοιτώντα τη στρατηγική τη ε, Κομισιόν για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, προβλέπεται να δοθεί ρόλο κλειδί στο ΕΦΣΙ, στο Ταμείο Γιούγκερ, για τι στρατηγικέ επενδύσει. Ποια είναι η εμπειρία σας μέχρι στιγμής ε, όσον αφορά τη χρήση αυτού του Ταμείου για τις υποδομές. Και μετά ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, υποθέσεις που εσείς γνωρίζετε και όπου έχουν ληφθεί μεγάλες ε, χρηματοδοτήσεις αλλά χρειάζονται υποστήριξη από την Ευρώπη και μετά μιλάμε για περιστρατηγικής κατά την άποψή σας λείπει κάτι από τη στρατηγική. Σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε στη μείωση των εκπομπών. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Κόχ. Ευχαριστώ και εγώ ένα ερώτημα για τον κύριο Ζούτα. Όπω είπε και ο συνάδελφο Βάντεκαπ, με εντυπωσίασε αυτό το, ε, ο αριθμό των 500 ε, δισεκατομμύριων ευρώ κατέτος εξωτερικό κόστο δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το ύψος του κόστους, όσο η κοστοαποδοτικότητα. Σίγουρα θα έχετε εξετάσει και την κοστοαποδοτικότητα, τη σχέση δηλαδή ωφέλους κόστους. Μπορείτε να μας πείτε δύο στοιχεία για αυτά. Ο κύριος Ρικέ, ένα... έχω ένα, πρόβλημα, ένα ερώτημα για τον κύριο Ζωνάρα, αλλά έχω και άλλα. Ε, ε, ε, αυτή τη στιγμή οι έρευνες αφορούν τους θερμικούς κινητήρες, ε, στα συμβατικά αερίου, ε, βιοκαύσιμα υγρά, βιοκαύσιμα αερίου, ε, διάφορα ευρυδικά, ευρυδικοί κινητήρες, μπαταρίες υδρογόνου. Δεν νομίζετε ότι όλοι αυτός, αυτός ο κατακρεματισμός, αν θέλετε, που μπορεί να οδηγήσει όλους σε μια μετάβαση πιο ομαλή, μήπως τελικά δεν έχουμε βρει όμως τη σωστή οδό μήπως δεν έχουμε μια κατεύθυνση πραγματικά προς το μέλλον. Θέλω να είμαι αισιόδοξο βέβαια στο τέλος. Καταφέραμε ε, να καταργήσουμε τις ατμομηχανές ε, άνθρακα. Ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ. τώρα βλέπω τους εμπειρογνώμονες εδώ. Είναι πολλές οι ερωτήσεις ε, για τα 500 δις και το εξωτερικό κόστος, ε, για το θέμα των χρηστών. πολλά ερωτήματα δεν θα τα αναφέρω όλα για να μην χάνουμε και χρόνο. Έχετε αγαπητοί πυρογνώμονες, δύο λεπτά. Ο καθένας, ναι ο καθένας, εντάξει. Δεν θα σας μοιράσουμε δύο λεπτά σε όλους. Βλέπω ότι παρακολουθείτε, ακόμα και αν είναι αργά όλοι παρακολουθείτε, πολύ ωραία. Εντάξει, παρακαλώ. Εδώ δεξιά. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για να απαντήσω στο, θέμα του στο ερώτημα του κ. Βαν Κάμπ. Η διαφορά ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι, συγγνώμη, δεξιά, δεξιά από του εμπειρογνώμους, από την υπηρεσία πρώτα, την υπηρεσία περιβάλλοντο και μετά. Ναι, δεν είπα ότι ήθελα να δώσω το λόγο στον Ακριανό. Παρακαλώ. Δεν είχα καταλάβει ότι αφορούσε εμένα ε, το ερώτημα. Δεν ξέρω αν τέθηκε ένα ερώτημα μόνο σε μένα, δεν, δεν ήμουν σίγουρος. Ακούστε, να πω κι εγώ δύο λόγια. Γίνεται μεγάλος λόγος για την αποδοτική χρήση της ενέργειας. Ε, ε όταν μιλάμε για το ποιε λύσεις πρέπει να βρεθούν, ε, ε είναι θέμα απόδοση. Βεβαίω πρέπει να επενδύσουμε σε νέα καύσιμα. Ε, είναι μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το είδαμε και στο γράφημα. Το να μειώσουμε δηλαδή την εκπομπή δεξιού του άνθρακα σε αυτό το επίπεδο θα χρειαστεί να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά και άλλα. Πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία. Όταν μιλάμε λοιπόν για μετάβαση, πρέπει να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές στην κοινωνία που θα καταστήσουν εφικτή αυτή τη μετάβαση λέμε στην έκθεση ε, ότι είναι και άλλοι τομείς. έτσι. Δεν είναι μόνο οι μεταφορές. Υπάρχουν μεταφορές, υπάρχει χρήση της γης, υπάρχει μηχανία, υπάρχει γεωργία, υπάρχει ο τουρισμός. Όλα αυτά κάνουν τη διαφορά τελικά όταν μιλάμε για τις εκπομπές ε, και τις μεταφορές τις εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών. Διότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση από αλλού. Ήθελα να αναφερθώ έτσι στο συστημικό, συστημική πτυχή του ζητήματος. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στη συμπεριφορά του κόσμου, διότι είναι προφανής η διασύνδεση των μεταφορών με την, εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Το θέμα είναι όμως ε, ποιες είναι, οι ποιες είναι διάφοροι τρόποι μεταφοράς που, που χρειάζεται η, οικονομία μας, ε, ποια χρειαζόμαστε λιγότερο. Σε επίπεδο αστικό υπάρχουν ορισμένα προφανή παραδείγματα νομίζω. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο διπλανός σας έχει το λόγο τώρα. Ναι, ακούστηκαν πολλά ερωτήματα που απευθύνθηκαν ιδίω σε μένα, ιδίω όσον αφορά την ε, μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Δεν μπορώ να σας τα πω. Ε, ε, υπάρχει εδώ και 20-30 χρόνια μια μεθοδολογία ε, για τον υπολογισμό του ε, εξωτερικού κόστους. Ε, σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα ατυχήματα και άλλες επιπτώσεις που προκαλούνται από διάφορους τομείς. Ή σε, αυτούς, σε αυτούς τους δείκτες και τα κριτήρια πολλές φορές προστίθεται και νέα, όπως είναι για παράδειγμα οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα στη δική μας περίπτωση. Ε, είπατε ότι θέλετε για στοιχεία για την ακρίβεια των, των ε, πληροφορίες για την ακρίβεια των στοιχείων μας ε, και παρατηρώ ότι όποτε αποκαλύπτονται ή δημοσιεύονται τέτοια στοιχεία ε, αλλάζει και ο χαρακτήρας της συζήτησης γιατί αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ότι κανένας τελικά τρόπος μεταφοράς δεν ανταποκρίνεται ή δεν αντισταθμίζει το, τη βλάβη που προκαλεί στο περιβάλλον. Ε, φυσικά δεν μπορεί ε, να συγκρίνει κανείς την αποδοτικότητα και το κόστος άμεσα με αναλογία ένα προς ένα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η τάση είναι σαφής και από αυτήν την τάση προκύπτει και η ανάγκη ε, η, ο κλάδος των μεταφορών να αναλάβει τις δικές του ευθύνες αλλά και το κόστος. Ε, για τα όσα προκαλεί. Ε, ίσως ε, μια τέτοια ανάλυση βεβαίως θα μπορούσαμε να την ε, επιχειρήσουμε και ίσως να αποδειχθεί και πολύτιμη. Όσον αφορά τις, τα μέτρα νομίζω που, που, που είναι αναγκαία για τη μετάβαση από τον έναν τρόπο μεταφοράς στον άλλον νομίζω ότι καλταλληλότερος θα ήταν ο ελφετός συνάδελφός μου να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Βαν Κάμπ, ε, αν συγκρίνουμε τη ΣΥΠΑ με την Ευρώπη, κάνατε μια έκκληση να γίνει σύγκριση μεταξύ ρεαλισμού και αισιοδοξία. Ε, η ρεαλιστική πτυχή είναι ότι η αγορά στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη ε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Διαφορετικέ είναι οι νομικέ απαιτήσει για τα φορτηγά στη ΣΥΠΑ και διαφορετικέ στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο τα φορτηγά έχουν και διαφορετική εμφάνιση. Το δικό δίκτυο επίσης είναι διαφορετικό στι ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ωφέλιμου βάρους, μεταξύ ε, απαιτήσεων ε, εμπορευμάτων στα ρημουλκούμενα. Αν δείτε λοιπόν την κατανάλωση καυσίμου, ε, ένα χιλιόμετρο, τα ευρωπαϊκά φορτηγά εκπέμπουν 60% λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα από τα αμερικανικά σήμερα ακόμη και χωρίς να έχουμε πρότυπα για τα φορτηγά στην Ευρώπη. Αν δείτε τι έχουν κάνει οι κατασκευαστές φορτηγών, τι έχουν επιτύχει την τελευταία πενταετία, θα αντιληφθείτε ότι ε, έχουν μειώσει την ε, κατανάλωση καυσίμου κατά 8% κατά μέσο όρο. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι σε τελική ανάλυση η κατανάλωση καυσίμου ε, μειώνει και το κόστος του μεταφορέου το 1 τρίτο από ό,τι κατάλαβα και θα σας πει ο συναδελφός μου εδώ στα δεξιά, το 1 τρίτο του κόστους των μεταφορών σχετίζεται με την κατανάλωση καυσίμου. Υπάρχει λοιπόν και εμπορικό κίνητρο εδώ ε, ώστε οι κατασκευαστές να παράγουν ε, ε, φορτηγά χαμηλότερης κατανάλωσης. Γιατί αυτό ζητούν και οι πελάτες μας. Αυτή είναι η αιτία. Δεύτερον, Όσον αφορά τις επενδύσεις σε εναλλακτικά συστήματα κίνησης, ε, το ερώτημα του κ. Ντεμεσμάκερ. Άμα δείτε εκεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, σε διάφορες περιοχές, ουσιαστικά δεν πρέπει να δείτε τις διάφορες περιοχές όπου υπάρχουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αρκεί να δείτε ποιος έχει αιτηθεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας και, ε, και, πού και, ποιο, και θα δείτε ότι πολλοί κόσμος έχει πάρει διπλώματα ευρεσιτεχνία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και αν δείτε μετά τα συστήματα κίνηση. αν δείτε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα παγκοσμίω, η Κίνα ηγείται, είναι μεγάλη αγορά φυσικά, η Ευρώπη είναι αριθμό 2 και η ΕΠΑ είναι αριθμό 3. Απλά για να το γνωρίζετε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μέντια, έχετε εσεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομο. Πολλά ερωτήματα έγιναν και μπορεί να απαντήσω και γραπτό στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι η πρόταση του κ. Άρχουγκ για συγκρισιμότητα και καλύτερη διαφάνεια είναι εξαιρετικά καλοδεχούμενη. Ο κλάδο δεν έχει τίποτα να κρύψει. Όμω πρέπει να συγκρίνουμε μήλα με μήλα και όχι με πορτοκάλια. Πρέπει να δούμε το θέμα των οδικών μεταφορών και γενικότερα. Η ιδιωτική ε, μεταφορά, ε, επαγγελματικέ υπηρεσίε, η επαγγελματική υπηρεσία στον οδικό ε, τομέα πρέπει να ε, συγκριθεί με τους άλλους τρόπους πάλι στον τομέα των πραγματικών υπηρεσιών όμως, μπορούμε να, να χτίσουμε δρόμους προς τις πλωτές οδούς και μπορούμε να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη χρήση του κάθε τρόπου μεταφοράς. Κύριε Λόγκριν, νομίζω ότι στη Σουηδία, κύριε Λόγκριν, αυτό το παράδειγμα που δώσατε, εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Εάν δεν μπορεί κάποιος ε, να οδηγήσει ένα λεωφορείο με τρόπο ε, ο οποίο να είναι υποφελής. Δεν καταλαβαίνω πώ μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί ένα τέτοιο λεωφορείο. Πρέπει οπότε έχει νόημα να αλλάζει το, το μοντέλο. Όμω, συμφωνώ με τον κύριο Βαν Κάμπ, δεν χρειαζόμαστε ε, λιγότερε οδού. οδούς, χρειαζόμαστε καλύτερες οδούς. 70% ε, εξυπηρετούμε εμεί ε, αυξάνεται η επαγγελματική μεταφορά, οπότε πρέπει να δούμε πώς αυτό θα γίνει καλύτερα και πιο έξυπνα σε ό,τι αφορά τώρα τα περαιτέρω σχόλια που ακούστηκαν. Ο κύριος Κράμερ, σας ευχαριστώ διότι επιβεβαιώσατε την πρόταση που κάναμε στην αρχή ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και τις αλλαγές της συμπεριφορά του κάθε κλάδου και ο κλάδος τον οποίο προσωπώ εγώ το πιστεύει αυτό. Τέλος, μας παρεμποδίζουν, μας δημιουργούν προβλήματα οι διαφορετικές διασυνοριακές, εθνικέ εθνικές πολιτικές μάλλον. Εμείς ε, το μας εμπόριο μας είναι διασυνοριακό. Ακούω προηγουμένως ε, ε, στην, στο Ρότερνταμ απαγορεύεται το, το, τα λεωφορεία diesel το 2020, από το 2020 και μετά. Έχουμε επίσης την οδηγία για την εναλλακτική χρήση που λέει το 2025 ε, θα πρέπει να αλλάξουμε, αλλά δεν, δεν ταιριάζουν όλα αυτά μεταξύ τους. Πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα και ε, όταν παίρνουμε δύο οχήματα, κυρία Ντέλη, πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι κάνει το καθένα από τα οχήματα αυτά και αυτό ε, απαιτεί διαφορετική τεχνολογία και διαφορετική μορφή ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούς έχει το λόγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για τις εκπομπές κύκλου ζωής, ένα θέμα που τέθηκε από πολλούς. Ε, υπάρχουν ε, στοιχεία για όλους τους τρόπους μεταφορών όσον αφορά τις εκπομπές κύκλου ζωής, τόσο για, τα, για τις δημόσιες όσο και τις επαγγελματικές όσο και τις ε, ιδιωτικές μεταφορές και δείχνουν όλα τα στοιχεία ότι ο σιδηρόδρομος είναι ο πλέον φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς. Ε, έχει πάρα πολύ μικρές επιπτώσεις. Σε ορισμένε περιπτώσει, βεβαίω, όλα αυτά εξαρτώνται από πολλού παράγοντες. Μιλώ πάντοτε για το μέσο όρο και την τάση. Για... Όσον αφορά την ε, προώθηση των ε, διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών, συμφωνώ ότι πράγματι ε, χρειάζονται επενδύσεις για να διευκολυνθεί η ε, μεταφορά ε, ε, των τρέιλερ των ρουμολικούμενων πάνω στα, στους σιδηρόδρομους, στους σειρμούς. Χρειάζεται οδική υποδομή και επενδύσεις στον τομέα αυτών προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η μεταφορά. Και ταυτόχρονα χρειάζεται να δημιουργηθούν και προσφορές αντίστοιχες για να γίνουν όλα αυτά. Πώς θα γίνουν αυτά? Πώς θα πείσουμε τον κόσμο να κάνει τη μετάβαση προς τους σιδηρόδρομους, βεβαίως χρειάζονται κίνητρα. Αυτό που κάνουμε στην ε, Ελβετία ε, σχετίζεται βεβαίως με, την, ε, με μια ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική, ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμη η μετάβαση στους σιδηροδρόμους για τις επενδύσεις. Μπορώ να σας πω τη λύση που έχουμε βρει στην Ελβετία με, έχουμε μία, εδώ και ένα χρόνο, ένα ταμείο ε, ε, υποδομών, το οποίο καλύπτει τη συντήρηση και την επέκταση των σιδηροδρόμων που χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές. Είχαμε και μια ψηφοφορία φέτος και δημιουργήθηκε ένα αντίστοιχο ταμείο και για τις οδικές μεταφορές για τους δρόμους. Και με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται και χρήματα, αλλά δίνεται και η δυνατότητα να σχεδιαστεί ε, με ανθεκτικό προς το μέλλον τρόπο η οδική και η σιδηροδρομική μεταφορά. Ωραία, το λόγο έχει ο κ. Νοβάτσκι είναι σημείωσα τις τρεις ερωτήσεις Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις φιλοδοξίες της αεροπορίας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση λόγω της αύξησης ε, της κίνησης, ε, της ενέργειας κίνησης. Στόχος ε, είναι να μειώσουμε το, τις εκπομπές μέχρι το 2050, πώς θα το επιτύχουμε. Έχουμε μια σειρά θεμέλιων λίθων, θέλουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό στην Ευρώπη, αλλά όπως ανέφερα ε, πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε την καινοτομία. Και όπως είπα εδώ στην Ευρώπη έχουμε το Team Sky Project, ε, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα, 4 δισεκατομμυρίων ευρώ επί πενταετίας και χρηματοδοτείται και από τον κλάδο. Είναι σημαντικό λοιπόν αλλά αν συγκρίνετε τι γίνεται αλλού, εμείς αν δείτε τι επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, ε, πόσα εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα αντιληφθείτε πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση. και ζητάμε από τους υπευθύνους χάρη πολιτικής να βοηθήσουν αυτά τα σημαντικά προβλήματα έρευνας. Σημείωσα μία ερώτηση που αφορά τι αεροπορικέ μεταφορέ σε σχέση με τι σιδηροδρομικέ. Ε, έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό πριν από 20 χρόνια. Η δημιουργία τη ενιαία αγορά αερομεταφορών που άλλαξε τελείω ε, τον κλάδο των αερομεταφορών. Ε, οδήγησε σε έντονο ανταγωνισμό. Χθε προετοιμάζοντα τη συζήτηση αυτή θυμήθηκα μια υπόθεση ε, που αναφέρουν συχνά οι περιβαλλοντικές ε, ΜΚΟ, ε, πώ είναι ένα ταξίδι μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνη. Ένα σιδηροδρομικό εισιτήριο από τη Μαδρίτη στη Βαρκελόνη υπάρχει μόνο μία εταιρεία ουσιαστικά. Γιατί η αγορά δεν είναι ακόμα ανοιχτή στις σιδηροδρομικές μεταφορές εντός της Ισπανίας. Ωστόσο, αν ψάξετε να βρείτε μια εταιρεια ουσιαστικα γιατι η αγορα δεν ειναι ακομα ανοιχτη στι σιδηροδρομικες μεταφορε εντο της ισπανια ωστοσο αν ψαξετε να βρειτε μια πτηση θα βρείτε πέντε αεροπορικές εταιρείες για την ίδια γραμμή. Τρεις ισπανικές, μια πορτογαλική ε, και μια νορβηγική. Με εντελώ διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, ευθυνέ, ε, ε, κλασικές κτλ. Οπότε ε, δεν μας εκπλήσει ότι στα μονοπόλια υπάρχουν υψηλέ τιμέ ενώ στις ε, ε, καταστάσεις υψηλού ανταγωνισμού υπάρχουν χαμηλές τιμέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ναι, σας ευχαριστώ. Να επανέλθω πρώτα στο θέμα, στο ερώτημα του κύριου Βαντεγκάμπ. Ακούστε, για τα παλαιά πλοία. Μπορεί να έχουμε ένα πολύ παλιό πλοίο με ένα νέο κινητήρα. Αλλά και με τον παλιό κινητήρα ε, δεν σημαίνει ότι ε, τα πάμε καλύτερα με τον νέο κινητήρα. Αυτό έχουμε βρει δυστυχώς με τις μετρήσεις μας ε, και ας είναι παράδοξο. Κάνουμε λοιπόν προσπάθειες για να δούμε ποιες είναι οι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και δεν είναι πάντα ίδια τα αποτελέσματα με αυτά που αναμένει κανείς σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Βεβαίως εμείς ε, θέλουμε να υπάρξει υποστήριξη από το Κοινοβούλιο ε, διότι και εμείς υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται για ένα καθαρό τρόπο μεταφοράς, ε, να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα ε, και να μοχλέσουμε χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από τον ιδιωτικό τομέα. Συζητούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και νομίζω ότι η υποστήριξή σα ε, εδώ θα ήταν εξαιρετικά καλοδεχούμενη, διότι υπάρχει τεράστια βούληση από το κλάδο να προχωρήσει. Τώρα, πιο κάτω, το ερώτημα της κυρίας Μάισνερ. για την αλλαγή των τρόπων μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ούτε με την αγορά των προϊόντων χίδινου, των κοντέινερ. Των κοντέινερ η, διαφορά, η δυσκολία είναι να μπορέσουμε να διεισδύσουμε σε νέες αγορές υπηρετικές και ήδη ξεκινάμε ε, με την κατάρτιση ε, πολύ λίγα μπλέγονται όταν κάποιος ε, μαθαίνει για αυτά τα πράγματα, ε, για τις εσωτερικές πρωτές οδού. Δηλαδή φτάνει κάποιος στον κλάδο αυτόν και δεν έχει ιδέα, δεν έχει καταρτιστεί, δεν έχει επιμορφωθεί. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια λοιπόν στον τομέα τον εκπαιδευτικό να περιλαμβάνονται και οι εσωτερικές πρωτές οδοί. Κάτι άλλο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι η αναθεώρηση της οδηγίας RIS ε, είναι το ETS των ιστορικών πλωτών ε, οδών αυτό. Ε, όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με, τους, με τις συνθήκες κυκλοφορίας, ε, το να γνωρίζουμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το εμπορευμά μου, πότε θα φτάσει. Αυτά σε συνολικό επίπεδο θα θέλαμε να είναι διαθέσιμα ε, για τον κλάδο να είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί στις εσωτερικές πλήτες οδού ε, θέλουμε να έχουμε πλήρη πλοία, να είναι γεμάτα, διότι αυτό είναι ε, και πιο συμφέρον οικονομικά αλλά και οικολογικά. Χρειαζόμαστε όμως την ανθεώρηση της οδηγίας, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και βεβαίως χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές και στην διασύνδεση και αυτό για την ώρα δεν έχει λειτουργήσει στα πλαίσια του ΕΦΣΥ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να πω για τον κύριο Βάντεκα ότι ε, γνωρίζουμε ότι η στρατηγική του IMO πρέπει να είναι φιλόδοξη. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς θα τα καταφέρουμε αυτό. Γνωρίζοντα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΑΕΜΟ, το καλύτερο είναι να αποφύγουμε την πόλωση μεταξύ ε, ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν θα πρέπει να πάμε και να θέσουμε τελεσίγραφα ε, για να πιέσουμε καταστάσεις οι οποίες μπορεί και να ε, εκπυρσοκροτήσουν στο τέλος σε μια αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε. Όσον αφορά το ερώτημα του, της κυρίας Μάισνερ, την ε, αλλαγή των τρόπων μεταφορών, αυτό αφορά και τις, ε, τις, ε, τις ε, ναυτιλιακές μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα καθήκον για την ναυτιλία, που είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, γιατί είμαστε ο μοναδικός τρόπος μεταφοράς που δεν λειτουργεί ακόμα στο πλαίσιο ενιαίας αγοράς. Νομίζω ότι με την υποστήριξή σας εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα ε, και να προχωρήσουμε μπροστά. Όσον αφορά τις ε, εγκαταστάσεις λιμένων, δεν έχω συγκεκριμένο κατάλογο των λιμένων, αλλά υπάρχει ε, διάλογος μεταξύ των αυτιλιακών εταιριών και των λιμένων, ιδίως μεταξύ των εταιριών κρουαζιέρας, προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα, να λυθούν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Και εδώ υπάρχει ένας διάλογος μέσα του οποίου μπορούν να αναπτυχθούν τα, ε, ε, προβλήματα. Ε, ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνολογία για τη μείωση των θιούχων εκπομπών, αλλά υπάρχει εκεί μια αντιφατικότητα μεταξύ των εκπομπών των θιούχων της, της για τις θιούχες εκπομπές και της οδηγίας για την ποιότητα του νερού. Ε, υπάρχει εδώ ένα θέμα νομικής ε, ε, αβεβαιότητας ώστε να γνωρίζουν οι εταιρείε ότι αν επενδύσουν στο Scrabble τότε πραγματικά θα μπορέσουν και να το αξιοποιήσουν. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν αναδυθεί. Λοιπόν, κλείνοντας λόγο στον εισηγητή. Πολύ σύντομα να... Ευχαριστώ ε, όλους ε, τους ομιλητές. Νομίζω ότι στην έκθεση θα έχουμε την ευκαιρία να ε, ε, επεξεργαστούμε ζητήματα οριζόντια που σχετίζονται με την επιμελητία, με την συμπεριφορά. Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα εξετάσουμε οριζόντια και μετά βεβαίως από εκεί και πέρα θα δούμε και κάθετα τον κάθε κλάδο, τον κάθε τομέα, τον κάθε τρόπο μεταφράσης προκειμένου να καταγράψουμε όλες τις διάφορες εξελίξεις που υπάρχουν. Ένα στοιχείο που προκύπτει και από τη σημερινή συζήτηση και που σχετίζεται και με τα όσα είπε ο κύριος Βαντεκάμπ είναι ε, η ανάγκη να εξευρεθεί μια ισορροπία. Γιατί αν δει κανείς ε, την, τον επίγοντα χαρακτήρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και την ανάγκη όλοι οι τομείς να κάνουν ε, τα δικά τους βήματα προς την κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, εκεί θα πρέπει να βρεθεί η ισορροπία. Και νομίζω ότι θα ήθελα να πω μάλλον στον κύριο Βαντεκόμ ότι εδώ το δίπολο δεν είναι αισιοδοξία ρεαλισμός, γιατί οι στόχοι που έχει θέσει το Παρίσι είναι ρεαλιστική. Πρόκειται για την αποφυγή της ε, κλιματικής αλλαγής. Μιλούμε δηλαδή για, έναν, για ένα δίπολο ρεαλισμού και ρεαλισμού ταυτόχρονα. Στις 31 ε, Απριλίου, ε, στις 30 Απριλίου μάλλον θα έχουμε ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης ε, που θα αποτελέσει και την έναρξη της συζήτησης και του έργου αυτού. Euh, Να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο γιατί πραγματικά ήσασταν στο ύψος των περιστάσεων, το αναμέναμε βέβαια, σας χρειαζόμαστε ακόμα όμως, μόλις αρχίζουν οι συζητήσεις, οι εργασίες στην Επιτροπή μας θα συνεχιστούν σε ό,τι αφορά την κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές και ο εισηγητής μας, οποίος τον οποίο ευχαριστώ και πάλι διότι προείδρευσε και του πάνελ, είναι ένα θέμα λοιπόν που μόλις τώρα αρχίζουμε να εξετάζουμε, είμαστε ακόμα μακριά από τους στόχους που έχουν τεθεί. Πάνε πολύ γρήγορα τα πράγματα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Έτσι λοιπόν οι καθαρές μεταφορές, ε, είτε μιλάμε για τις οδικές μεταφορές, τις θαλάσσιες τις αερομεταφορές, ε, είμαστε ακόμα μακριά. Υπάρχει ήδη μόχλευση πάντως. Ε, εγώ που ασχολούμαι με τη βιώσιμη κινητικότητα χαίρομαι που ε, οι έξυπνες πόλεις, ε, τα τοπικά, πολεδομικά προχωρούν. Η το Μάλμο αυτή η Σουηδική πόλη πριν από δύο μέρες έλαβε το βραβείο των ΣΝΙΦΣ, της, το, το βραβείο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά την αστική πολεοδομία. Έγινε αναφορά προηγουμένως στην Ευρωσήμα. Ε, υπάρχει το σχέδιο Juncker για να περάσουμε σε τρόπους μεταφοράς που έχουν τρεις πομπές, ε, τους ποταμούς, ε, τα διάφορα, διάφορες μορφές μεταφοράς στις, της σύνθετες. Θα πρέπει στον τομέα της αυτοκινητομηχανίας και εκεί ε, να συνοδεύσουμε την όλη διαδικασία. δεν πρέπει να έχουμε τον κλάδο απέναντι στον νομοθέτη. Ε, έχουμε τις ίδιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Ε, βεβαίως ε, έχουμε, υπάρχουν και κάποιες ε, εκθέσεις και ελπίζω να πάμε προς μια πραγματική επαναβιομηχανοποίηση ε, του τομέα της Ε, Μιλάμε για 13 εκατομμύρια εργαζόμενους, έτσι, οπότε πολλά διακύβευαν εδώ. Καλή τύχη λοιπόν στον κύριο Μπασεκού που είναι ο σκιώδης εγγύης για το θέμα αυτό. Ελπίζω να σταθούμε στο ύψος, στο ύψος τώρα του διακυβεύματος, έτσι, για τον πλανήτη, για την υγεία των πολιτών. Μιλάμε για μόλυνση, ε, αλλά μιλάμε και για έναν οικονομικό ε, κλάδο εντό του οποίου κινούμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε νομίζω να ε, χειροκροτήσουμε και τους ειδικού αλλά και τους εισηγητές ε, που πραγματικά θα δουλέψουν σκληρά για το πλαίσιο αυτή τη φιλόδοξή ονομοδότηση. Ε, ne partez pas, ne partez pas. Μη φεύγετε όμως, μη φεύγετε. Συνεχίζουμε. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous voulez saluer nos Λοιπόν, αν θέλετε να αποχαιρετήσετε τους ομιλητές, παρακαλώ εκτός αιθούσης. Alors, je le répète, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous... Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κύριε Ερμπάς, λέει η πρόεδρος. Κύριε Τύρι Νοβάτσκι, παρακαλώ συνεχίστε έξω τη συζήτηση. Πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ. À très bientôt. Merci les experts. À très bientôt. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σημείο 9 της μέση διάταξη Προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσει προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ θα υποβληθεί. Δίνουν το λόγο στον κύριο Κιθ Τέιλορ. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και στους διάφορους εισηγητές και θα μπορέσουμε επίσης να καλέσουμε την Κομισιόν να πάρει το λόγο και να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Ο κύριος Τέιλορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συγκεκριτές για την επικοδομητική σου συμμετοχή και για την υπομονή τους. Έγιναν πολλές ε, συζητήσεις και υπήρξαν και κάποιες διαφωνίες βασικά. Εκτιμώ ιδιαίτερα την αφοσίωσή τους ε, στο στόχο του να επιτύχουμε κάποια συμβιβαστική λύση για κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Δυστυχώς οι γνώμες δίστανται σε τέτοιο βαθμό γεγονός που μας οδήγησε να ζητήσουμε αναστολή της ψηφοφορίας ε, ε, για την γνωμοδότηση αυτή για άλλες δύο εβδομάδες, ώστε να επιτευχθεί κάποιο συμβιβασμός. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Ε, ωστόσο, σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή συζητάμε την εξέταση τροπολογιών, ενώ δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα οι συμβιβαστικές για πολλά σημεία έχουμε συμφωνία συμπεριλαμβανομένου του θέματος ε, βελτίωσης της νομοθετικής συνοχής. Ωστόσο, απομένουν διάφορα πολιτικά σημεία ανεπίλητα. Το σημαντικότερο είναι το ζήτημα του οικοδομημένου περιβάλλοντος, ε, των, ε, των υπηρεσιών μεταφορών και προϊόντων εντό δομημένων περιβαλλόντων. Πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την οδηγία και οι εταιρείε μεταφορών θα πρέπει να λάβουν μια δίκαιη και σωστή υποδομή, ε, προθεσμία, υποδο, προθεσμία συγγνώμη, ε, όσον αφορά την προσβασιμότητα για ανθρώπους μειωμένη κινητικότητας. Ε, Αμφιβάλλω αν θα συμφωνήσουμε με πολλούς συναδέλφους. Απομένουν πολλές διαπραγματεύσεις ε, ακόμα για το, να δούμε το, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθούν όλα αυτά. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό και για την προσβασιμότητα στα μηχανήματα πληρωμών, ελέγχου και στα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης. Οι περισσότερες ε, ομάδες έχουν συμφωνήσει ότι όλα αυτά τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι απολύτως προσπελάσιμα. αλλά πρέπει να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες τώρα όσον αφορά τις προθεσμίες υλοποίηση και τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Και τέλος, ένα συμβιβασμό για το κατά πόσο τουριστικές υπηρεσίες όπως ε, υπηρεσίες διαμονής και ε, σύντησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο της, ε, της οδηγίας και αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση. Οπότε έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο μέχρι στιγμής στις αρχικές μας συζητήσεις. το σημαντικό για αυτό το νομοθέτημα είναι ότι θα διασφαλίσει ε, κάποια αυτονομία σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα και είναι πολύ σημαντικό θέμα. Απομένουν πολλά να γίνουν ε, στο διαπραγματευτικό μέτωπο. Ε, θα έχουμε μια συνάντηση σκιωδών την επόμενη εβδομάδα και στο Στρασβουργό και θα το ψηφίσουμε στις 11 Απριλίου στην Επιτροπή. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό αποδεκτό για όλες τις ομάδες. Ε, πάντα υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Ε, α, ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο μιλητής και έχει φύγει η Πρόεδρος. Να αντικαθιστώ εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα επανέλθει. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στον σκιώδη συγκητή, στους σκιώδης πρώτα ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κρίς ε, Τέιλερ θερμότατα για το έργο του. Ως συνειδητής της διακοινοβουλευτικής ομάδας για τις αναπηρίες πριν από πολλά χρόνια ε, θεωρώ ε, πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα που αφορούν τους, ε, τα άτομα με αναπηρίες. Και γι' αυτό ε, αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά να ε, αποφέρουμε απτά αποτελέσματα για τους ανθρώπους αυτούς. Άρα, αυτά αφορούν οπωσδήποτε το δομημένο περιβάλλον, τον τουρισμό, την πρόσβαση στις παραλίες, στις ακτές, και τα ζητήματα της εργασίας. Εμείς ως ΕΛΚ είχαμε ε, ορισμένα ε, προβλήματα και ορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με την αρχική πρόταση ε, της Κομισιόν για τον τουρισμό. Εδώ δεν υπάρχει αρμοδιότητας. Οι επιπτώσεις δε θα είναι τρελές αν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να μετασκευαστούν όλα τα παλάτια για παράδειγμα που μάλιστα είναι και διατηρητέα κτίρια προκειμένου να είναι προσβάσιμα από όλους τους τουρίστες. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άλλα μέσα, για παράδειγμα η ψηφιοποίηση. Στις αστικές συγκοινωνίες ε, είναι τόσο περίπλοκο θέμα που δεν, μπορούν, που δεν μπορεί να ρυθμιστεί ούτε καν στο πλαίσιο μιας ε, οδηγίας για τις ε, αστικές συγκοινωνίες αυτές καθεαυτές. Αυτό που ελπίζω ε, είναι στην ε, από εδώ και πέρα συζήτηση να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να ξαναεπανεξετάσουμε ε, τις διατάξεις που αφορούν τις μεταφορές και το δομημένο περιβάλλον και να ελέγξουμε μήπως θα έπρεπε να συντάξουμε ξεχωριστή εισήγηση αντί να εντάξουμε τα πάντα σε αυτήν εδώ την ε, εισήγηση ε, και στη συγκεκριμένη οδηγία. Άλλωστε, πολλές από τις αρμοδιότητες εξακολουθούν να εμπίπτουν σε εθνική ε, να είναι εθνικής, πολλές αρμοδιότητες εξακολουθούν να είναι εθνικές. Γι' αυτό και αυτό που χρειάζεται εμείς να κάνουμε είναι να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και τι μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ε, ε, μη ρεαλιστικές ε, προτάσεις. Αντιθέτως, αυτό που πρέπει να είναι στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε ένα ρεαλιστικό κείμενο το οποίο θα μπορεί να την χάνει της υποστήριξης της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Τραν. Εγώ προς το παρόν δεν πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κείμενο. Παρ' αυτά μπορώ να συμφωνήσω και εγώ με την αναβολή της ψηφοφορίας, της ε, οδηγίας. Ε, δεσμεύομαι να συνεχίσουμε την ε, συνεργασία μας με τον εισηγητή και θα ακολουθήσουμε αυτήν την οδό και στο διάστημα από εδώ και πέρα. Ο κύριος Έρτογκ, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους σκιώδεις. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Ζένα Λόουερ λόγω του ότι συμμετέχει σε συνάντηση σκιωδών στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Σας διαβάζω λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειές του να εξευρεθούν συμβιβασμοί μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων. Εμείς υποστηρίζουμε τις περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες. Αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, ε, ώστε να καλύπτονται και οι αστικές συγκοινωνίες, ε, τα συστήματα ενημέρωσης και πληρωμών. Ε, επίσης υποστηρίζουμε τον συμβασμό ε, για την αποφυγή επικάλυψης νομοθετημάτων. Θα πρέπει η οδηγία αυτή να καλύπτει ζητήματα που δεν καλύπτονται νομοθετικά μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ε, όπου αυτό δεν ισχύει, θα πρέπει να ισχύει η ε, ευρωπαϊκή πράξη για τα άτομα με αναπηρίες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ε, εμπίπτουν οι υπηρεσίες για το δομημένο περιβάλλον στο πεδίο εφαρμογής αυτού της οδηγίας. Είναι κρίσιμη σημασία για τα άτομα με αναπηρίες όταν αποφασίζουν να ε, επιλέξουν ε, τρόπους ε, μεταφοράς. Υπάρχουν στο παράρτημα 1 διάφορες απαιτήσεις για τις κινητές εφαρμογές, τα συστήματα πληρωμής και ε, νομίζω, ότι θα πρέπει ε, το παράρτημα αυτό να ε, επικεντρώνεται σε, και σε μηχανήματα πληρωμής ή ακύρωσης εισιτηρίων, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ακόμα. Επίσης υποστηρίζουμε την ανάγκη ένταξης των εφαρμογών κινητών συσκευών στον τομέα των μεταφορών. Ελπίζω να τύχουν υποστήριξη αυτές οι προτάσεις μου και θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τον εισηγητή και τους, τους σκιώδεις εισηγητές για την συνεργασία τους και ελπίζω να καταφέρουμε εν ευθέτω χρόνο να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις ώστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή ΙΜΚΟ να ε, λάβει υπόψη της τις ε, δικές μας συστάσεις. Αυτά από την σκιώδη μας, την κυρία Σιναλόερ και ε, θα ήθελα να επαναλάβω εδώ την αφοσίωσή της ώστε να ξεπεραστούν τα, τα όποια προβλήματα έχουν εμφανιστεί στη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Τελίτσκα. Ε, Δυστυχώ η συνάδελφος αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής της ε, αποστολής παρατηρητών στο Ανατολικό Τιμόρ. Ε, οπότε θα, θα αναφέρω εγώ κάποια στοιχεία που ήθελε να αναφέρει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε καταρχήν ποιο είναι ο στόχο εδώ. Ο στόχο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφωθεί με τι νέε υποχρεώσει που απορρέουν από την ε, Σύμβαση των Μένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Η κυρία Μπιλμπάου θεωρεί ότι μόνο μία ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα δημιουργεί το κατάλληλο νομικό περιβάλλον και, που δεν θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμού. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. Δεύτερον, ίσω να πρέπει να με αυτό, η κυρία Μπιλμπάου εκτιμά ιδιαίτερα ε, το κείμενο του κυρίου Τέιλορ, αλλά για μια σειρά ζητήματα ε, δύσκολα η ομάδα των σχεδόν εισηγητών είναι κάπως ε, ε διαιρεμένη. Ε, θεωρεί ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση. Ε, ίσως θα ήταν πρόημο να το αναβάλουμε. Ε, θα γίνει κάθε προσπάθεια πάντως από την κυρία Μπιλμπάγκα να φτάσουμε σε μια κοινώ αποδεκτή λύση, σε μια κοινώ αποδεκτή συμφωνία. Ένα σημαντικό ζήτημα εδώ είναι ότι πρέπει να δούμε αυτή την νομοθετική πρόταση ως κάτι που έχει να συμπληρώσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα δικαιώματα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και με αναπηρία όταν ταξιδεύουν με, τους διάφορα, με τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Ε, θεωρεί λοιπόν η συνάδελφος ότι αυτή η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν οι απαιτήσει προσβασιμότητας δεν καλύπτονται από καμία άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, να αποφύγουμε και τα κενά. Ε, σε ό,τι αφορά τα ευαίσθητα ζητήματα τώρα, ε, το περιβάλλον. Υπάρχουν εδώ δύο σχολές, ε, βέβαια, ε, στην Επιτροπή μας, ε, αλλά και στην ομάδα των σχεδόν εισηγητών. όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα δύο στρατόπεδα. Η κυρία Φρανσίσκο Μπιλμπάο ε, λέει ότι έχουμε ε, δύο ισορροπημένες ε, ομάδες σε επίπεδο σχετισμού, σχετισμού δυνάμεων. Κάποιοι προτιμούν την αρχική πρόταση να συμπεριλάβουμε το περιβάλλον αλλά εθελοντικά. Ας το εξετάσει αυτό ο εισηγητής μου πως αυτή είναι μια λύση ε, να βάλουμε το building environment δηλαδή εδώ, αλλά εθελοντικά. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τουρισμό, ε, θέλω να επενθυμίσεις και ως εισηγήτρια ότι η συμπερίληψη του τουρισμού σε καμιά περίπτωση δεν αντιβαίνει το άρθρο 195 της συνθήκης που ε, θέτει το θέμα της πολιτικής τουρισμού στην δημοκρατία των κρατών μελών, αλλά οι υπηρεσίες αυτές ε, που συνδέονται με τον τουρισμό καλύπτονται και από την οδηγία, τουρισμού, την οδηγία υπηρεσιών συγγνώμη, 123 Οπότε αυτομάτως έχουμε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Δύο ακόμα σχόλια. Και όλη η συγγήτρια μου ζήτησε να υπογραμμίσω ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση αυτή η οδηγία να οδηγήσει σε διοικητικό άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τις νέες επιχειρήσεις λέει ότι το βάρος, το άχθος θα πρέπει να είναι αναλογικό. Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε δυσανάλογο άχθος. Γι' αυτό λοιπόν προτιμά να υπάρχει μια νέα προϋπόθεση που θα λαμβάνει υπόψη τις εναλλακτικές, ε, τις δωρεάν εναλλακτικές ε, που ε, παρέχουν η παροχή υπηρεσιών μεταφορά. Υπάρχουν δηλαδή εναλλακτικέ. Ε, και τελευταίο σχόλιο. Η σκέψη εισηγήτρια θέλει να υπενθυμίσει ότι αλλού, όπω στι ΗΠΑ αλλά και σε άλλε χώρε στην Νότια Αμερική, η προσβασιμότητα σε υπηρεσίε και προϊόντα είναι ήδη πραγματικότητα και είναι ε, εκ των νουκ άνευ για να μπορέσει κάποιο να συμμετάσχει στο εμπόριο, στην αγορά τη συγκεκριμένη. Πρέπει λοιπόν τα προϊόντα μα, οι υπηρεσίε μα, να καταστούν πιο προσβάσιμα και έτσι να καταστούν και πιο ελκυστικά. Είναι ένα στοιχείο ε, που ε, έχει και μια εμπορική χρειά και αυτό είναι που μου ζήτησε ε, η συγκίτρια να τονίσω ω τελευταίο. Νομίζω δεν ξέχασα τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τιλίτσκα. Ο επόμενο ομιλητή. Α, δεν θέλετε το λόγο. Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πλασέντσια να πάρει το λόγο λοιπόν για να μας δώσει κάποια στοιχεία. Okay, very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να επιτύχουμε μια ε, συμφωνία σύμφωνα και με τις απόψεις της Επιτροπής αυτής. Να επισημάνω δύο πράγματα ε, όσον αφορά τα όσα ακούσαμε σήμερα. η προσεκτική μέρημνα με την οποία η Επιτροπή έλαβε υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία και συμπληρώνει αυτά που υπάρχουν ήδη, αποφεύγοντας ε, τις επικαλύψεις. Δεύτερον, ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να παρασχεθεί προσβασιμότητα και να διευκρινίσουμε ότι αυτό δεν αφορά την ύπαρξη εναλλακτικών όταν τα πράγματα δεν είναι προσπελάσιμα. Επικεντρώνεται η οδηγία στο πώς θα επιτευχθεί η προσβασιμότητα με τρόπο συνεκτικό και εναρμονισμένο σε ολοκλήρη την Ένωση. Αυτά είναι τα δύο σημεία που θα ήθελα να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Τέλορ. Αν έχετε σχόλια. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Για μένα και για τους πράσινους και για πολλούς ε, από τους σκιώδεις η οδηγία αυτή θα πρέπει να αφορά την επέκταση των υπηρεσιών μεταφορών και των προϊόντων ώστε να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι εντός της ενιαίας αγοράς. Αυτός ο στόχος υπάρχει, αυτή η φιλοδοξία υπάρχει. Ακούστηκε και ε, το γεγονός ότι πρόκειται για μια ε, αμοιβαία αποφελή διαδικασία. Το να βελτιώσουμε λοιπόν τις μεταφορές και τις υπηρεσίες για λίγους τελικά θα καταλήξει στο να τις βελτιώσει για το σύνολο. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Η ψηφοφορία λοιπόν δεν θα γίνει αύριο. Αλλά στις 11, έχει αναβληθεί για τις 11 Απριλίου. Θα ήθελα απλά να πω ότι δεν θα μπορέσει να αναβληθεί ξανά, διότι αυτό αλλάζει όλε τι εργασίε τη Επιτροπή. Δεν γίνεται αυτό, κάποια στιγμή πρέπει να ψηφίσουμε. Εγώ έκανα τώρα μια εξαίρεση για την έκθεση αυτό, ε, αλλά δεν πρόκειται να την ξανα... επαναλάβω. Οι προθεσμίες πρέπει να τηρούνται, διότι υπάρχουν και οι άλλε επιτροπέ ε, που αναμένουν τι εκθέσει για γνωμοδοτήσει. Δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε το νομοθετικό έργο από την Επιτροπή μα. Συνεχίζουμε τώρα τι εργασίε μα και θα ζητήσω, επειδή θα συνεχίσουμε και κλεισμένο των θυρών, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να κοπεί η άμεση μετάδοση και να καλέσω το κοινό να εγκαταλείψει την αίθουσα. Κυρίως το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Παρακαλούμε να χωρίστε.